Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας ακρόαση. Θα θέλαμε να αρχίσουμε. Σας παρακαλώ, ησυχία. Χαιρόμαστε για την ανθρώπινη προσέλευση. Ζητώ συγγνώμη, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές θέσεις μέσα αυτή την αίθουσα. Κάποιοι θα χρειαστεί να μην όρθιοι. Ε, θα έρθουν κάποια καθίσματα, αλλά όχι πολλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Να καλωσορίσω ε, και το ακροατήριό όμως που μας παρακολουθεί από το διαδίκτυο. Επί της διαδικασίας ζητώ συγγνώμη που αργοπορήσαμε, αλλά είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση για την οδηγία περί προστασία των καταναλωτών και θα ήθελα να απευθυνθώ στου ε, βουλευτέ τη επιτροπής μα για να ανακοινώσω το εξή Αύριο το πρωί 10 η ώρα ε, θα, θα συζητήσουμε ένα επιπρόσθετο σημείο ούτως ώστε να εγκριθεί το τελικό κείμενο για την οδηγία προστασίας των καταναλωτών. Οι πολιτικές ομάδες ε, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα το υπερψηφίσουν. Αύριο το πρωί λοιπόν θα γίνει μια πάρα πολύ σημαντική συνεδρία. Είναι σημαντικό όλοι οι βουλευτές να προσέλθουν αύριο το πρωί και μετά το επόμενο βήμα είναι η Ολομέλεια, η μήνυ Ολομέλεια στις Βρυξέλλες για τελική έγκριση. Λοιπόν, ενιαία αγορά τώρα και ε, τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση. Αυτό είναι το θέμα της ακρόασής μας. Ε, συνάδελφος Σάλντε ήταν εισηγήτρια για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, για το θέμα αυτό στο παρελθόν. Είχε αυτή η έκθεση κέρια σημασία διότι προσανατόλισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ακολούθησε μια εκτεταμένη μελέτη την ε, αρχική πράσινη βίβλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίζω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει έρθει πολλά και στην Επιτροπή μας και έχει καλύψει βασικά, πολύ βασικά ζητήματα και τώρα είσαστε αρμόδια για τα τυχερά παιχνίδια. Να, μια νέα πρόκληση για σας. Σας καλωσορίζω και πάλι. Καλωσορίζω επίσης τον Γιώργεν Κρόιτσμαν, από τους φιλελευθέρους, ε, ε, σκληρέ εργαζόμενος συντονιστής, αλλά και εισηγητής για τη δεύτερη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τα τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά, που έχει ιδιαίτερη σημασία διότι προχωρά εκ παραλίλου και επωφελείται από τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για το ζήτημα. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν για τη συμμετοχή όλων. Θα κάνουμε κάποιες εγωικές παρατηρήσεις ε, για να πλαισιώσουμε το υποσυζήτηση θέμα. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και κάποιους από τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριο Διό πρέπει να αποχωρήσει νωρί, το ξέρω και αν δεν έχουν πρόβλημα οι σκιώδεις θα αντιστρέψουμε τη σειρά παρέμβασή τους. Κατόπιν θα ακούσουμε σύντομα σχόλια από του σκιώδεις εισηγητές αν το επιθυμούν. Ουδάλλως οι σκιώδεις εισηγητές ούτως ή άλλως ε, θα μπορέσουν και στη συνέχεια της συζήτησης ε, να παρέμβουν όποτε το επιθυμούν διότι θέλουμε να, λίγο μετά τις 4 να αρχίσουμε να ακούμε τις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων. Γιώργεν Κρόιτσμαν, ε, θα σου δώσω αμέσω το λόγο, δίχω περαιτέρω καθεστήριση, Παρακαλώ για να αρχίσει τη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Όπως ξέρετε όλοι, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε ένα μοσαϊκό ρυθμίσεων σε κάποιες χώρες, π.χ. στη Γερμανία απαγορεύονται τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, αλλού όπως στη Μάλτα, τη Μεγάλη Βρετανία έχουν πιο φιλελεύθερο καθεστώς. Επίσης υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, Δανία, Ιταλία που επιτρέπουν τα παιχνίδια στο διαδίκτυο αλλά με αστηρή αδειοδότηση. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι πάρα πολλές αποφάσεις του ΔΕΚ και οι διαδικασίες επί παραβάση που έχει κινήσει η Κομισιόν. Παρά λοιπόν την διαφορετική κατάσταση είναι διαθέσιμος ο τζόγος σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω και της μαύρης αγοράς και του ότι βασίζεται σε ε, υπεράκτιες έδρες. Οπότε η κατάσταση δεν θέλω να την ικανοποιητική αλλά ούτε και ιδιαίτερα δραματική. Χαίρομαι επίσης πέρα από τους συναδέλφους για το ότι ανέλαβε μια πρωτοβουλία και η Κομισιόν για μια πράσινη βίβλη για αυτό το σημαντικό θέμα. Μου είπαν πως η Κομισιόν στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων αναμένει πάρα πολλές παρεμβάσεις, κάτι το οποίο τονίζει τη σημασία αυτού του θέματος, ε, κάτι το οποίο καθίσταται φανερό και μέσα στην αίθουσα οι προτεραιότητες της έκθεσής μου. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων. Ξέρετε πως εδώ πέρα ισχύει η αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή πρώτα απ' όλα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη ε, για το αν θέλουν να ανοίξουν τις αγορές τους στο τζόγο, στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει λοιπόν ε, να αποφασίσει να μην επιτρέψει κάτι δεν μπορεί να του το επιβάλλει η Ευρώπη. Αν όμω υπάρχει ε, άνοιγμα τη αγορά θα πρέπει να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία χωρίς διακρίσεις. Αυτό σημαίνει παραδείγματο χάρη πως ε, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός αδειών για κάθε ε, ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία θα πληρεί τις προδιαγραφές. Επίσης, δεν ε, επιτρέπεται παραδείγματος χάρη να προσδιοριστεί πόσο σερβερ θα πρέπει να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι και οι ρυθμίσεις που ισχύουν και κατά την άποψή μου θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως για κάποιες πτυχές της ρύθμισης αγοράς πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν δεν υπάρχει πλειοψηφία γι' αυτό τότε τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία το θέλουν στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας όπως ακριβώς έγινε και για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, να κάνουν μια κοινή ρύθμιση. Αλλά τονίζω πως ε, τα κράτη-μέλη σε ένα τέτοιο σύστημα θα εξακολουθούν να έχουν την κυριαρχία όσον αφορά την απόδοση των αδειών. Βεβαίως ε, θα πρέπει το σύστημα να διαμορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν ε, κίνητρα για να ζητήσει κανείς άδεια για να περιοριστεί η μαύρη αγορά. Δεύτερον, η προστασία των παιχτών, να καταπολεμηθεί δηλαδή και η εξάρτηση και ο τζόγος ε, των ανηλίκων και το οργανωμένο έγκλημα. Η Κομισιόν το έχει τονίσει πάρα πολύ αυτό το θέμα στην Πράσινη Βίβλο και βεβαίως θα κάνω και εγώ προτάσεις στην ε, έκθεσή μου. Και Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω ιδέες και τη συναδέλφου Σάλντε Μόζε. Θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές έτσι ώστε πανευρωπαϊκώς να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Τέλος, ο σύνδεσμος μεταξύ στοιχημάτων και αθλητισμού είναι πάρα πολύ σημαντικός καθώς κατά κανόνα στα κράτη-μέλη αυτά τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών. Äh, από την άλλη όμως ε, για να μπορέσει να γίνει αυτό και στο μέλλον θα πρέπει μέσω της αρχής της επικουρικότητας να διατηρούν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να δίνουν άδειε ε, και να καθορίζουν την χρήση. Πέρα από αυτό βεβαίως χαίρομαι για τα σχόλια των συναδέλφων σχεδόν εισηγητών των άλλων ομάδων με τους οποίους συναντηθήκαμε για να προετοιμάσουμε αυτή την ακρόαση και καλέσαμε βέβαια όλους τους παρευρισκόμενους για να έχουμε ένα ευρύ φάσμα απόψεων ε, από όλα τα κράτη-μέλη. Πάλι για το χρονοδιάγραμμα Ξέρετε πως ε, μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε το σχέδιο, τροπολογής μέχρι τις 20 Ιουλίου, ψηφοφορία με την εβδομάδα της 19ης ε, Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή και Ολομέλεια στον, ε, στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο. Λοιπόν, να δούμε ποιε κοιόδε θα ήθελαν ίσω συντομία το λόγο πριν να αρχίσουμε την ακρόαση. Και πρέπει να φύγει, επομένω να του δώσουμε καταρχήν το λόγο και κατόπιν οι υπόλοιποι σκιώδε. Μπορείτε να μου κάνετε νόημα αν θέλετε το λόγο. Λοιπόν, ας ε, ξεκινήσουμε, κύριος Δεόν, κύριε Φόξ, κυρία Ρούλα κτλ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για το ότι θα πρέπει να φύγω, αλλά σε λίγο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχουμε ψηφοφορίες. Βεβαίω ο συνάδελφος ε, κ. Τριανταφυλίδης θα παραμείνει εδώ πέρα και εκπροσωπείται άρα η ομάδα μας. Πρέπει να πω πως είναι πολύ ζωντανό το αντικείμενο, βλέπω, φαίνεται αυτό και από τον αριθμό των ανθρώπων που ήρθαν και ήθελαν να έρθουν. Και ξέρετε πως ε, ούτως ή άλλως αν δει κανείς μόνο για τα έσοδα του Λότος ένα έτος μιλάμε για 80 δισεκατομμύρια. Είναι για μια τεράστια επιχείρηση αλλά ελπίζω να αντιληφθούμε πως δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή οικονομική ε, δραστηριότητα. Αναφέρθηκαν οι πτυχές της δικαιοσύνης ε, και χαίρομαι που τα ανέφερε αυτά ο κύριος Κρότσμαν καθώς και το ότι υπάρχει ζήτημα επικουρικότητας. Βεβαίω στη πράξη υπάρχουν ε, προβλήματα. Αν δούμε και τη χώρα μου παραδείγματο χάρη την Ολλανδία υπάρχει σαφές πρόβλημα χειρισμού της κατάστασης και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τις ε, κρατικές ε, αρχές. Στο πλαίσιο του, του τζόγου και του στοιχήματος καθώς επεκτείνονται αυτές οι εταιρείε γενικότερα στον τομέα της, ε, της ψυχαγωγίας. Γιατί εντάξει θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την επικουρικότητα αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το κράτος μετά μπορεί να δημιουργεί ε, έτσι απλά μονοπόλια. Και πρέπει οπωσδήποτε να τα συζητήσουμε αυτά, να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι λειτουργίες του κράτους. Αλλά όπως σας είπα για εμάς δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη οικονομική δραστηριότητα, πρέπει να υπάρχει προστασία για την εξάρτηση από τον τζόγο και να δούμε τις πρακτικές οι οποίες υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κύριος Φόξ. Ευχαριστώ την Κομισιόν που παρουσίασε αυτή την πράσινη βίβλο, γιατί ε, πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν σέβονται τους κανόνες αγοράς και δημιουργούν ουσιαστικά εμπόδια στην ελευθερία της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών και αυτό δεν μπορούμε να το, να το επιτρέψουμε να συνεχίζεται. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα σε ό,τι αφορά τα υπεύθυνα τυχερά παιχνίδια και να προστατεύσουμε τους ευπαθείς καταναλωτές. Νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει από τον κλάδο σε αυτό το τομέα, σε συνεργασία ε, με της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα για ένα νομικό πλαίσιο. Η πράσινη βίβλος που εκπονήθηκε από την Κομισιόν δεν ήταν το πιο ισχυρό έγγραφο της Κομισιόν που έχω δει μέχρι σήμερα. Δεν έθεσε μια ξεκάθαρη στρατηγική πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να θαρρύνω το Κοινοβούλιο να είναι τολμηρό και να δώσει απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις που η Κομισιόν φαίνεται να θέλει να απαντήσει, να, να αποφύγει με συγχωρείτε. Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους συνσηγητέ να είναι θεραλέοι και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Κομισιόν για να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα δημιουργήσει θέσει εργασία και καινοτομία, αλλά και θα επιφέρει και έσοδα φορολογικά στα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία δεν κατάλαβα. νομίζω ότι θα ήταν οι άλλες ομάδες. Δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Θέλω να ακούσω πώς θα κυλήσει η ακρόαση. Νομίζω πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από όταν καταλήξαμε σε μια κοινή θέση με την κυρία Σαλτεμόζα, αλλά είμαι ανοιχτή στο να μου αλλάξετε την άποψη. Ναι, και εμείς, και εμείς μπορούμε να το πούμε. Er Βασικά, δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε που ψηφίσαμε επί της έκθεσης ε, το Μάρτιο του 2009. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ελέγχουμε αυτά που υπόθηκαν δηλαδή είναι ουσιαστική η αρχή της επικορικότητας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίσουν πώς θέλουν να ρυθμίσουν αυτή την αγορά των τυχερών παιχνιδιών στην κάθε χώρα. Αλλά δεν υπάρχει βέβαια και καμία αμφιβολία ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε και τους καταναλωτές και τους ευπαθείς αλλά και τους ανηλίκους. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση αυτών των συγκεκριμένων θεμάτων. Επίσης πρέπει να δούμε αν ε, εφαρμόζουμε σωστά την νομοθεσία, μήπως μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να αναλυφθεί δράση κατά ε, όσων ε, κατέχουν παράνομα άδειες. Εγώ ανυπομονώ να ακούσω τους εμπειρογνώμονες εδώ σήμερα, να ακούσω τι είναι ουσιαστικό εδώ να πράξουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε και πεθερό λιγμών στα κράτη-μέλη και θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς την αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προστατεύσουμε ε, τους παίκτες, παύλα καταναλωτές. Ε, όταν ε, μιλάμε για τα τυχερά παιχνίδια, πάντοτε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλοί άνθρωποι παρευρίσκονται εδώ σήμερα, έχουμε αθρέο προσέλευση. Έτσι λοιπόν, ενυπομονώ να ακούσω όσα έχετε να πείτε. Ευχαριστώ και τέλος ο κ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Απηχώντας την παρέμβαση του εισηγητή και της κυρίας Σάλντε Μόζε, θα προσέθετα κι εγώ ότι επιχαίρουμε για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει επιτάπητος αυτό το ζήτημα ε, μέσα σε μια πιο χαλαρή ε, ήπια ατμόσφαιρα και άρα μπορούμε να εργαστούμε αποτελεσματικά. Πρώτον. Δεύτερον, ε, τα τυχερά παιχνίδια διαφέρουν από τις υπόλοιπες αγορές ε, και η υπηρεσία προσφοράς δηλαδή τυχερών παιχνιδιών διαφέρει από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Μιλήσαμε για προστιθ... ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η κυρία Σαλτεμόζε δίκιο έχει και μας μιλάει για την προστασία των καταναλωτών και κυρίως των ανηλίκων. Αλλά θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, σχετίζεται με την ίδια την ακαιρεότητα των τυχερών παιχνιδιών και αυτό συνδυάζεται με την προηγούμενη έκθεση. Δηλαδή, εκεί εξετάζεται την ακαιρεότητα των ε, τυχερών ε, ε, παιχνιδιών και είχατε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω όπως εισηγητής κάποια τέτοια στοιχεία που σχετίζονται ούτως ή άλλως με την επικουρικότητα. Εγώ θα μιλούσα μάλιστα για την δραστήρια επικουρικότητα, δηλαδή να επιδιώξουμε να βρούμε κοινά, ρεαλιστικά, τεχνικά κριτήρια ε, σχετικά με την αδειοδότηση παραδείγματο χάρη, ούτως ώστε να σημειωθεί η πρόοδο και να είναι ελκυστική η προσφορά, ε, η θεμητή προσφορά, ε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις δόλιες προσφορές ε, και να οικοδομήσουμε ένα μηχανισμό συνεργασίας ή τουλάχιστον βελτίστων πρακτικών. Δεύτερον, εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης στον τομέα αυτό. δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να συμμορφωθούν όλοι με την αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση. Επίση, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρώτο απολογισμό από το άνοιγμα των αγορών σε κάποια κράτη-μέλη. Πρώτον, πρώτα απ' όλα, μάλλον, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με του φορεί που προσφέρουν υπεράκτιε υπηρεσίε. Ε, το ανέφερε ο εισηγητή και νομίζω ότι τα περικατάχρηση τη εσωτερική αγορά ε, είναι ε, ζητήματα που πρέπει να μα απασχολήσουν πρωτίστω. Οπότε, ανακεφαλαίοντος, να πω, να ε, σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας, μη εφαρμογή της αρχής αμοιβαία αναγνώρισης και συνεργασία για να επιδιώξουμε μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, ευρωπαϊκά στοιχήματα παραδείγματο χάρη, ούτω ώστε τα έσοδα να διοχετεύονται όπως θα έπρεπε στην αγορά και οι αθλητικές ενώσεις να μπορέσουν να επιβιώσουν, όπως σωστά είπατε, και ταυτόχρονα να επεξεργαστούμε κοινά τεχνικά πρότυπα, χάρη στα οποία οι φορεί ε, εκμετάλλευσης, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς θα μπορέσουν να ε, υποβάλουν μια ενδιαφέρουσα νόμιμη, θεμητή προσφορά ε, και να υποφεληθούν οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ όλους. Ε, νομίζω ήταν ε, χρήσιμο να πλησιώσουμε τη συζήτηση με αυτές τις εναρκτήριες παρεμβάσεις και τώρα όσοι σας ακούν, όσοι σας βλέπουν γνωρίζουν ποια είναι η θέση των πολιτικών ομάδων, των συντονιστών των πολιτικών ομάδων για το θέμα αυτό. Είναι τα πρόσωπα κλειδιά πέρα από τον εισηγητή. Ας περάσουμε τώρα στο σημερινό πρόγραμμα των ειδικών προσκεκλημένων των εμπειρογνωμών, πιο συγκεκριμένα που έχουμε προσκαλέσει σήμερα και κατόπιν θα ακούσουμε με τι ερωτήσει των βουλευτών και τις απαντήσεις. Έχουμε μία σειρά εμπειρογνωμόνων ε, με ευρεία πραγματογνωμοσύνη σε πολλούς και διάφορους τομείς. Θα αρχίσουμε ε, ασχολούμενοι με την αγορά των τυχερών παιχνιδιών σε απευθεία σύνδεση και πώς μπορεί να ρυθμιστεί η αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατόπιν οι επαγγελματίες του κλάδου και όσοι εμπλέκονται με τις ρυθμιστικές διατάξεις ε, θα, μας, ε, θα τοποθετηθούν σχετικά με την ε, εξέταση ενός σχεδίου κανονισμού για τη ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών. Μετά θα ασχοληθούμε με την πλευρά των καταναλωτών. Υπάρχουν πολλοί ε, που έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα για τα κοινωνικά προβλήματα, το παθολογικό τζόγο, παραδείγματος χάρη ε, και ε, όλοι γνωρίζετε ότι παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ο τομέα των τεχειρών ε, παιχνιδιών και δεν μπορούν να γίνουν παραλληλισμοί ε, ούτε να αντιγράψουμε οι υφιστάμενες δημόσιες πολιτικές. Τέλος πάντων, ας μην μακρηγορώ γιατί έχουμε μια μεγάλη σειρά ομιλητών και πρέπει να ελέγχουμε αυστηρότατα το χρόνο. Θα χρονομετρούμε τους ομιλητές και αν υπερβείτε το χρόνο αγόρευση, θα αρχίσω συνοφριώντα τα φρύδια μου, κάνοντα γκριμάτε και μετά αν δεν υπακούσετε έχω και το σφυράκι. Ε, μέσα στους φακέλους έχετε ε, τα διάφορα έγγραφα και τις διαφάνειες ε, για τις παρουσιάσεις που ήταν διαθέσιμες ήδη εκ των προτέρων. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα ο κύριος Λόρι Κόρπι, που είναι ο νομικός διευθυντής και διευθυντής ερευνών του Gambling Compliance και έχει μεγάλη πραγματογνωμοσύνη στον ε, τομέα αυτό. Θα μας μιλήσει για 10 λεπτά και θα ακολουθήσει ο κύριος Φίλιπ ε, Φλέμινγκ που εργάζεται στην Fleming Partners ε, και έχει εκτεταμένη εμπειρία ε, ως προς ε, τους νόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλούς και διάφορους τομείς. Έχει ξανάρθει στην Επιτροπή μας όχι μόνο για τα τυχερά παιχνίδια και για άλλα θέματα και επίσης είναι ακαδημαϊκός και ερευνητής στον τομέα αυτό. Ο χρόνος αγόρευσης θα οριστεί στα 10 λεπτά. Κύριε Κόρπη. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες διαφάνειες. Καλό θα ήταν να τις δούμε και στην οθόνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μπορώ να σας δώσω ορισμένε πληροφορίες. Εργάζομαι για τον Gamble Compliance εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και θέλω να ε, δώσω κάποιες πληροφορίες εναντί ε, της πράσινης βιβλίου σε σχέση με το πώς μοιάζει η αγορά στα τυχερά, των τυχερών παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα αναφερθώ σε ορισμένο ρυθμιστικό τρόπο, αλλά θα δούμε δεδομένα πολύ την Ευρώπη. Επόμενη διαφάνεια. για να ξεκινήσουμε. Βλέπετε εδώ στο χάρτη αυτό Ξέρουμε ότι πολλά κρατημέλη έχουν ένα είδος ρύθμισης ε, για τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και λίγες χώρες ρητός απαγορεύουν τη δραστηριότητα αυτή. Υπάρχουν ε, ορισμένες γκρίζες αγορές εκεί, δεν ε, υπάρχει νομοθεσία στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε περαιτέρω κατανομή της ε, γκρίζας ζώνης. Εδώ βλέπετε στις ρυθμισμένες αγορές ε, στην Ευρώπη υπάρχουν ε, κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ του μονοπωλίου λίγο πολύ και ανοιχτής αγοράς, αποκλειστικής άδειας και ανοιχτής αγοράς και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ε, ουσιαστικά ότι συνοδεύει την πράσινη βίβλο, έρχεται η πράσινη βίβλο στη στιγμή που υπάρχει δραστηριότητα στα κράτη-μέλη. Εδώ βλέπετε τα κράτη-μέλη στα οποία λαμβάνει η χώρα κάποια δραστηριότητα σε σχέση με το επιγραμμικό ε, με τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια η Ισπανία πρόσφατα ψήφισε νομοθεσία ε, και ε, η Δανία επίσης έλαβε κάποια μέτρα ενώ η Φιλανδία έγραψε τα μονοπωλιά της σε νομοθεσία ε, και η Γερμανία σήμερα απαγορεύει τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και βλέπετε εδώ ότι φτάνουμε μέχρι, από δυτικά μέχρι ανατολικά την Κύπρο. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και την Ιταλία που επέκτηνε φέτο τα επιγραμμικά προϊόντα της για να συμπεριλάβει το καζίνο και το πόκερ ή τη Γαλλία η οποία συμπεριέλαβε με ρήτρα θεώρησε στην ομοθεσία ε, για τα τυχερά παιχνίδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυναμική εξέλιξη στον τομέα τη στιγμή που δημοσιεύει δημοσιεύεται η πράσινη βίβλος. Τώρα να δούμε την επόμενη διαφάνεια η ερώτηση είναι τι μαθαίνουμε αν δούμε τα προϊόντα. Ε, τα κράτη-μέλη υπάρχουν συγκεκριμένα νομικά πλαίσια και όλα τα προϊόντα ρυθμίζονται σε συγκεκριμένα στάδια. Το αθλητικό στοίχημα επιτρέπεται συνήθως επιγραμμικά και ακολουθούν τα προϊόντα λαχιοφόρου αγορά και στη συνέχεια το καζίνο και το πόκερ σε πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα κράτη-μέλη. Όμως ε, υπόκεινται σε αλλαγέ όλα αυτά. Αν δούμε την επόμενη διαφάνεια, ε, εδώ ε, τι μπορούμε να συμπεράνουμε για την αγορά βάση των δεδομένων. Νομίζω ότι η Πράσινη βίβλο ε, αποκάλυψε πολλά στην πρώτη υποσημείωσή τη όταν είπε ότι υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία. Αυτό είναι αλήθεια, καθώ μόνο η Ιταλία και η Γαλλία μηνιαίω ε, και τριμηναίω δημοσιεύουν ε, στατιστικά στοιχεία στο ίντερνετ για τα τυχερά παιχνίδια, αλλά είδη πηγών δεδομένων όπως μελέτες δεν είναι ε, διαθέσιμες σε όλες τα κρατημέλη. Έχουμε μία πρόχειρη δουλειά δεδομένων ε, επί των οποίων οι ερευνητές, ε, οι και οι εμπορευόμενοι έχουν πρόσβαση. Αν, να αν μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια, αν δείτε εδώ ορισμένα από τα διαθέσιμα στοιχεία, ε, η ΑΜΣ στην Ιταλία ε, ουσιαστικά μας έδειξε ορισμένα στοιχεία για το πώς ρυθμίζονται οι επιγραμμικές λειτουργίες ε, της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Εδώ βλέπετε και κάποια παιχνίδια δεξιοτήτων η Ιταλία επέκτηνε τη ρυθμισμένη αγορά της ε, για να συμπεριλάβει και τα παιχνίδια σε μετρητά και τα παιχνίδια καζίνο. Και καθώς ε, υπάρχει ισχυρή βάση θα μπορούν οι ε, νομοθέτες ε, να κρίνουν ποια επέκταση της αγοράς έχει γίνει αλλά και οι εμπορευόμενοι όταν θα σκεφτούν αν θα μπουν στην αγορά ή όχι. Η Ιταλία έχει πληθώρα συνόλου δεδομένων. Εδώ βλέπετε τους ενεργούς λογαριασμούς χρηστών από μήνα σε μήνα. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν ε, τους χαράκτε πολιτική να αξιολογήσουν ε, μια πολιτική ε, που έχει να κάνει με τη ρύθμιση των προσφορών. Επόμενη διαφάνεια, Γαλλία και η Γαλλία αρχίζει να παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία. Εδώ βλέπετε μια απεικόνηση των ρυθμισμένων προσφορών, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Βλέπετε το σχετικό μέγεθος των τομέων και αν δείτε το αθλητικό στοίχημα, βλέπετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το αθλητικό στοίχημα στην Γαλλία. Όλα αυτά είναι τα δεδομένα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την αξιολόγηση της αγοράς. Επόμενη διαφάνεια. Αλλά τι συμβαίνει με την ε, υπόλοιπη επιγραμμική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εδώ αγωνιζόμαστε να βρούμε δεδομένα όπως υπάρχουν για τη Γαλλία και την Ιταλία. Εδώ έχω παρουσιάσει κάποια διαθέσιμα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε ορισμένες χώρες σε σχέση με το μέγεθος, παραδείγματος χάρη, της ε, γκρι αγοράς της Ισπανίας ε, σύμφωνα με τα δεδομένα της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας ή του Ηνωμένου, της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιγραμμικοί εμπορευόμενοι και Επίσης έχουμε στοιχεία από Γερμανία και Σουηδία, δύο εκτιμήσεις σε σχέση με το σχετικό μέγεθος αυτής της ε, αγοράς τυχερών παιχνιδιών στις δύο αυτές χώρες. Εδώ ένας άλλος τομέας όπου έχουμε δεδομένα είναι να εξετάζουμε ε, κάποιες επιχειρήσεις. Εδώ βλέπετε στοιχεία για την Ισπανία και την Ελλάδα. Υπάρχουν αναδυόμενες αγορές ε, περίπου 250 εκατομμυρίων ε, καθαρών κερδών. Σε εσοδέτηση λοιπόν με αυτά τα πρόχειρα δεδομένα και με ορισμένες εκτιμήσεις δημιουργείται μια εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς ε, επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών. Αν φτάσουμε τώρα στο τέλος παρουσίασης μου, τι μπορούμε να πούμε για την αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των τυχερών παιχνιδιών. Πώς μοιάζει σήμερα. Πρόκειται για μια σειρά αγορών που κινούνται από μετά ρύθμιση και παραμένουν κατακαιρματισμένε. Πολλέ αγορέ κινούνται γρήγορα. Τώρα, ε, η πρόσβαση σε ε, αξιόπιστα δεδομένα ποτέ δεν ήταν πιο κριτική σημασία από εμπορική σκοπιά. Παραδείγματο χάρη, πολλά ε, δεδομένα βασίζονται τώρα σε φορολογική πολιτική ορισμένα αναφέρονται στα έσοδα από το αθλητικό στοίχημα ε, και βλέπουμε όμως ότι μειώνονται τα επίσημα έσοδα γιατί ε, διωγγώνεται τα στοιχήματα στη μαύρη αγορά. Ε, εδώ εμείς θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν υπάρχει αντίθεση μεταξύ Ιταλίας, Βελγίου και Δανίας παραδείγματος χάρη με τα μεικτά έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια, τι πληρώνουν οι παίκτες και με την ε, Γαλλία και τη Γερμανία παραδείγματος χάρη αλλά το σίγουρο είναι ότι χωρίς αξιόπιστα δεδομένα ε, δεν θα είναι δυνατόν να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Ίσως να ήμουν θαραλέος ή ανόητος, αλλά ε, όταν ε, μου ανατέθηκε ε, αυτή η παρουσίαση εγώ προσπάθησα να σας παρουσιάσω τα στοιχεία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ που, δεχτή, που πας, σεβαστήκατε και το χρόνο. Νομίζω ότι η έκκλησή σας ε, για τα αξιόπιστα αυτά δεδομένα είναι κάτι που είδαμε και από την έκθεση ε, του κυρίου Κρόιτσμαν. Αλλά όταν θα έχουμε περισσότερα δεδομένα ε, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε. Φυσικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε βοηθούν τη συζήτησή μας. Ο κύριος Βλέμινγκ τώρα για 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι όλο που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να σχολιάσω αυτό το συναρπαστικό ζήτημα τη ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Ταυτόχρονα βέβαια συνιστά και πρόκληση. Το Πανεπιστήμιο τη ε, Λουβά ε, μου ζήτησε το ίδιο και χρειάστηκα ώρε για να παρουσιάσω το θέμα. Οπότε θα ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά έχω 10 λεπτά στη διάθεσή μου και θα περάσω γρήγορα τι διαφάνειε. Περάστε στην επόμενη ήδη παρακαλώ. Σε αυτή την παρουσίαση θα ήθελα να σχολιάσω ε, μία σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από την ε, νομολογία. Η όλη συζήτηση για την αμοιβαία αναγνώριση, η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, σχετικά με το αν χρειάζεται περιοριστική νομοθεσία ε, ή αν αρκεί η εθνική νομοθεσία, διοδότηση και τέλος το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των διοργανωτών των αθλητικών συναντήσεων. Επόμενη διαφάνεια. Εν είδη εισαγωγή να σας πω ότι η νομολογία ακόμη δεν είναι αποκρισταλωμένη παρότι έχουμε πολυάριθμες ε, ε, υποθέσεις ε, για τις οποίες έχει εκδώσει απόφαση από το 1994 και μετά το δικαστήριο. Εκρεμούν πάρα πολλές υποθέσεις κατά τη διάρκεια της ακρόασης και σε σχέση με την γνωστή Ιταλική υπόθεση και μια άλλη γαλλική υπόθεση, μια Αυστριακή υπόθεση απασχολούν την δημόσια γνώμη. Η αυστριακή υπόθεση μόλις κοινοποιήθηκε στα κράτη-μέλη. Δεν έχει λήξει λοιπόν η συζήτηση περί του δικαστηρίου. Επόμενο στοιχείο, επί σειρά ετών γινόταν συζήτηση σχετικά με το αν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί η αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση για τα τυχερά παιχνίδια, ε, βασιζόμενη σε μια άδεια που έχει εκδοθεί από ένα κράτο μέλο, ένα φορέα εκμετάλλευση θα μπορούσε ιδανικά να λειτουργήσει άλλα κράτη-μέλη. Το 99, στην υπόθεση Λάρα τη Φινλανδία, το δικαστήριο ε, τοποθετήθηκε και είπε ότι όταν επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να υιοθετούν δική του εθνική πολιτική, ε, σεβόμενη την πολιτική κάποιου άλλου κράτου μέλου έχουν ε, τη διακριτική ευκαιρία να αποφασίσουν ε, αν μπορούν ε, να δραστηριοποιηθούν στην επικράτειά του οι φορεί εκμετάλλευση και για ποιο είδο τυχερών παιχνιδιών. Ε, πρώτη φορά εκδόθη απόφαση ε, στην υπόθεση Λίγα Πορτογκέζα de Football, η, ε, Ευρωπαϊκή, η Πορτογαλική Λίγα Ποδοσφαίρου δηλαδή, όπου το δικαστήριο σαφέστατα είπε το εξή, το ότι ένα φορέα εκμετάλλευση προσφέρει νομίμω τι υπηρεσίε του σε κάποιο κράτο μέλο, αυτό δεν συνιστά επαρκή εγγύηση σχετικά με την πρόστασία των καταναλωτών σε ένα άλλο κράτο μέλο κατά τη απάτη. Η αρχή τη χώρα προέλευση δεν κατοχυρώνει ούτε την ακαιρεότητα ούτε τι επαγγελματικέ δεξιότητε του φορέα εκμετάλλευση και δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική και νόμιμη παροχή υπηρεσιών. Αυτά είπε το δικαστήριο και ξανασυζητήθηκε η απόφαση στην υπόθεση Λαντμπρο, όπου ε, επανέλαβε τη δήλωση ε, το δικαστήριο και μάλιστα ε, υπερθεμάτισε. Οπότε θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει ε, λυθεί, έχει επιληθεί από το δικαστήριο. Κατόπιν, ε, σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας, ε, από την πρώτη υπόθεση, το 1994 δηλαδή, θεώρησε το δικαστήριο ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι μια οικονομική δραστηριότητα ιδιαίτερης φύσης και ότι τα κράτη-μέλη έχουν ευρύ αρμοδιότητα να εκτιμήσουν τι είδους πολιτική θέλουν να ακολουθήσουν ε, στην επικράτειά τους. Και το δικαστήριο μίλησε για διακριτική ευχέρεια. Αυτή ε, τη φρασιολογία χρησιμοποίησε ε, στη νομική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μέλος έχει ευρύ αρμοδιότητα και περιορίζεται μόνο από την αυθαίρετη δράση ενός κράτου. Ε, και αυτό ε, προβλέπεται και στη συνθήκη, εφόσον προσπαθούμε να μελετήσουμε αυτό το θέμα στα πλαίσια τη συνθήκης. Λοιπόν, ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν ποιο είναι ο στόχο του, μπορούν να αποφασίσουν το επίπεδο τη προστασία των καταναλωτών που θέλουν να προσφέρουν, πώ θα διαφυλάξουν τη δημόσια τάξη, αν θα επιτρέψουν ή όχι και υπό ποιου όρου ε, ε, αυτά τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση και προφανέστατα οι κυρώσει ε, κατά των φορέων εκμετάλλευση που δεν έχουν την άδεια να προσφέρουν υπηρεσίε να διαφημίσουν στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτου μέλου. Συνεχίζουμε σε διάφορες υποθέσεις ε, το δικαστήριο είπε ότι ε, μία ε, προσέγγιση μονοπωλίου είναι πιο πρόσφορη σε σχέση με ένα σύστημα ανταγωνιστικής αδειοδότησης. Αρνείται το δικαστήριο την δυνατότητα στο κράτος μέλος να επιλέξει ή το ένα σύστημα ή το άλλο αλλά τίθεται κατά του μονοπωλίου διότι τίθεται ζήτημα εποπτείας σε σχέση με ένα ε, ανταγωνιστικό σύστημα ε, αδειοδότησης για τους αλλοδαπούς φορείς εκμετάλλευσης παρότι θα υπάγονται σε ένα σύστημα ε, εποπτείας. Λέω ξεκάθαρο, το δικαστήριο δεν απέκλεισε άλλες μεθόδους, απλώς εξέφρασε την προτίμησή του σε διάφορες αποφάσεις που έχει εκδώσει για αυτή την προσέγγιση. Επόμενο θέμα. Ε, η υπόθεση Ζινάτη, Βλαγγέλη, Φλαγκάτη ε, είναι άλλε υποθέσει όπου ετέθη το ζήτημα ε, των παιχνιδιών σε απευθεία σύνδεση, η υπόθεση Λίγκα Πορτογκέζα κτλ είναι υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με το θέμα. Και ποια ήταν η εκτίμηση ε, του δικαστηρίου ε, ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος ε, απάτηση και παραπλάνησης για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση σε σχέση με τα παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια και προέταξε τέσσερις λόγους που δεν ανέπτυξε, δεν εφήβρε το δικαστήριο, απλώς επανέλαβε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τη σχετική απόφαση όταν συζητήθηκε όταν ε, η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στη ΣΥΠΑ από την Αντίγκουα ε, μίλησε για το θέμα πρόσβασης, ε, το θέμα της συχνότητας, την ανωνυμότητα των φορέων εκμετάλλευσης και ρητά ανέφερε το δικαστήριο ότι το διαδίκτυο είναι απλώς ένας διάβλος και όχι ένα διαφορετικό είδος ε, τυχερού παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα αυτού αναγνώρισε το δικαστήριο ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν ε, την εφαρμογή των μονομερών περιοριστικών ε, όρων για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος διότι έχουν δημόσιο χαρακτήρα τα παιχνίδια σε επαυθείας σύνδεση και άρα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκή συμμόρφωση με τις εθνικές κείμενες διατάξεις. Περνάμε τώρα στον πυρήνα του ζητήματος Επίτροπος Μπαρνιέ στην δήλωση που έκανε πέρσι ήταν σαφής γιατί δεν τίθεται καν το ζήτημα η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ε, ο πυρήνας είναι η συνοχή της πολιτικής ε, και αυτό το θέμα το τόνισε και το δικαστήριο στην υπόθεση Ζινάτη και Γκαμπέλη. Οι περιοριστικές πολιτικές μπορούν να διατηρηθούν μόνο και μόνο, μόνο συγγνώμη, εάν συμβάλλουν ε, στην προστασία με συνεκτικό και συστηματικό τρόπο. Επόμενη διαφάνεια. Επικρατεί κάποια σύγχυση στα κράτη-μέλη μετά την υπόθεση Πλακάνικα, όπου το δικαστήριο τροποποίησε κατά τη δήλωσή του, προσθέτοντας ε, το δυναμικό ελέγχου της ε, επέκτασης. Ε, αυτό ακολούθησε και η υπόθεση Λάνσμπρουκ, δηλαδή μπορούν να έχουν περιοριστική πολιτική τα κράτη-μέλη και ενίοτε να ενισχύουν την καταπολέμηση της απάτης ή την καταπολέμηση των παρανόμων τυχερών παιχνιδιών ε, και το κράτος μέλος δικαιούται να έχει μια ελεγχόμενη επέκταση της εθνικής πολιτικής του ακόμη και να χρησιμοποιεί μονοπωλιακά μέσα ε, και μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφήμιση ή νέες μεθόδους διανομής. Ε, αφετέρου ήταν βέβαια σαφές στο δικαστήριο και σε διάφορες ε, υποθέσεις ε, μέχρι την, ε, τις πιο πρόσφατες άρχισε να υιοθετεί όλο και πιο περιοριστική πολιτική σε σχέση με τη διαφήμιση. Δηλαδή είναι σαφές ότι πρέπει να περιορίζεται στο ε, ελάχιστο απαραίτητο η διαφήμιση για τα εγκεκριμένα τυχερά παιχνίδια και ότι υπάρχουν τρόποι διαφήμισης κυρίως από ένα μονοπωλιακό φορέα που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την φυσική τάση του καταναλωτή να τυχερά παιχνίδια ή να ενισχύσουν τον εθισμό του. Ε, χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, πολύ λαμπερά χρώματα ε, για να ανακοινώσουν τα ιονή κέρδη ε, και άρα τονίζεται, υποδαβλίζεται η φυσική έξι των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο. Κατόπιν, ε, υπάρχουν πολλά πρότυπα, πολλά μοντέλα που μπορούν να συνεπάρξουν για τα τυχερά παιχνίδια, αλλά δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε μονοπόλιο για ε, τις λιγότερο επικίνδυνες μορφές ε, παιχνιδιών και να έχουμε ανοχή και ανοιχτή αγορά για τα, τις πλέον επικίνδυνες ε, μορφές τυχερών ε, παιχνιδιών. Σχετικά με την αδειοδότηση θα είμαι σύντομο. Ε, το δικαστήριο σαφέστατα μίλησε για το μοντέλο της διαφάνειας, της κατάλληλης διακριτικής συμπεριφοράς, διάκριση ανάμεσα στην μοναδική ενιαία αδειοδότηση ή την πολλαπλή αδειοδότηση. Επόμενη διαφάνεια, επόμενη. Είναι σαφές λοιπόν ότι ε, μπορείτε να έχετε μια περιορισμένη ε, διάρκεια και μια συγκεκριμένη μορφή. Τα βλέπετε στη διαφάνεια, δεν τα λέω κι εγώ. Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων ε, ετέθη το ζήτημα. Μόλις ε, συνειδητοποίησα ότι υπερβαίνω και το χρόνο αγόρευσή μου, στο συγγνώμη, ε, ε, οι διοργανωτέ των αθλητικών συναντήσεων έχουν πνευματικά δικαιώματα. Έχει γίνει η συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου σε διάφορες υποθέσεις. Υπάρχει και σχετική οδηγία. Συνεχίζεται η συζήτηση. Τώρα... Κλείνοντα, να πω ότι το δικαστήριο μα βοήθησε για να διευκρινίσουμε διάφορα ζητήματα. Φυσικά δεν έχουν ρυθμιστεί όλα ε, τα θέματα και άρα επικρατεί κάποια νομική ανασφάλεια. Σας Ευχαριστώ. Ξέρετε, δεν μπορώ να σα χειροκροτήσω γιατί έχω δεμένο το χέρι μου. Αλλιώ θα σα χειροκροτούσα. Γιατί ε, μπορέσατε να δείτε όλε τι υποθέσει ε, του δικαστηρίου και να κάνετε την ανασκόπηση μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Καταπληκτικό είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τώρα έχουμε προβλέψει χρόνο για ερωταπαντήσει. Ο κύριο Πιτέλα πρέπει να φύγει Ε, παρακαλώ κύριε Πιτέλα και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή και οποιοδήποτε άλλο θέλει να παρέμβει. Κύριο Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα καταρχήν ε, να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς ε, εισηγητές αλλά και τους συναδέλφους τους σκιώδεις ε, εισηγητές που ξεκίνησαν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φυσικά θα διαβάσω και όλα τα έγγραφα που μου έχουν χορηγηθεί. Θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή σας ε, ένα στοιχείο που αναφέρει η Κομισιόν ε, στην Πράσινη Βιβλίο ότι πάνω από το 85% των ενεργών ιστοσελίδων των γερών παιχνιδιών στην Ευρώπη λειτουργούν χωρίς άδεια. Είναι κάτι τρομακτικό. Μιλάμε για πάνω από το 85% χωρίς άδεια. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε λοιπόν μία διασυνοριακή αγορά η οποία κατά σε ένα μεγάλο βαθμό είναι παράνομη και ε, ενέχει πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους και για τους παίκτες αλλά και για τις κυβερνήσεις και για τους εμπορευομένους που φέρουν άδεια. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Νομίζω ότι μία από τις προτεραιότητες πρέπει να είναι με συγκεκριμένο τρόπο να προσδιορίσουμε τι εννοούμε με το παράνομο τζόγο και με το νόμιμα τυχερά παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχει δίκιο ε, συνάδελφος η οποία είπε ότι πρέπει να εγγυθούμε την αρχή της επικουρικότητα. Είναι σωστό. Αλλά έχουμε κοινέ αρχές επί των οποίων θα πρέπει να υπερισχύει για μια διασυνοριακή διάσταση. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει ανάγκη στα θέματα επί της όπως ε, αυτό το θέμα της νομιμότητας ε, ή του παράνομου χαρακτήρα των τυχερών παιχνιδιών να υπάρχει μια σαφής νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Jürgen κύριο κύριος Κορότσμαν, ο εισηγητής μας. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακούσαμε πως είχε λάβει κάποιες αποφάσεις. Μας τα είπε και ο κύριος Πιτέλα λόγω της μαύρης αγοράς και λοιπόν προβλημάτων και αν δεν υπάρχει καταγραφή δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε κιόλα. Οπότε ποιες ε, ευκαιρίες βλέπετε εσείς γιατί αφενός είναι σαφές πως τα κράτη-μέλη έχουν την αρχή της μπορούν να διατηρήσουν μονοπόλιο αν θέλουν. Δεν μπορούμε να τα εμποδίσουμε αλλά Νομίζω το είπε και ο πρώτος ομιλητής πως υπάρχει κινητικότητα όπως βλέπετε και στο χάρτη υπάρχουν άδειε ε, που δίδονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Βλέπετε δυνατότητα δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία επιθυμούν μια ρύθμιση. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Φλέμινγκ. Είπατε πως Παρ' όλα αυτά απαιτείται μια πολιτική λύση για νομική βεβαιότητα. Τι είδους πολιτική λύση. Μπορείτε να μας κάνετε κάποιες προτάσεις. Άλλος. Η κυρία Γκέπχαρτ, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αναφερθώ ακόμη μια φορά στο θέμα άδειες, ευρωπαϊκή αγορά. Ξέρετε όταν συζητήσαμε την ε, οδηγία υπηρεσιών πως είχε προβλεφθεί εκεί πέρα ως εμπορική υπηρεσία τα τυχερά παίγνια το οποίο εμείς το βγάλαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είπαμε πως δεν είναι μια απλή υπηρεσία χρειαζόμαστε ειδικέ διατάξεις είπαμε όμως τότε ή εγώ είχα πει τουλάχιστον πως η εξαίρεση από την οδηγία των υπηρεσιών δεν πρέπει να μας εμποδίσει να σκεφτούμε πως μπορούσαμε να δώσουμε ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα που προκύπτουν από το ίντερνετ. Γιατί δε, εκεί πέρα δεν υπάρχουν σύνορα. Και υπάρχει πάρα μια πάρα πολύ μεγάλη γκρίζα αγορά, πρόσβαση ε, και σε κράτη-μέλη στα οποία τελικά απαγορεύεται κάτι τέτοιο και έχουμε μια κοινή προσέγγιση και άρα το ερώτημά μου είναι ε, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε αφενός ε, να γίνει σεβαστή η επικουρικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα προστατευτούν και οι πολίτες και η οργανωμένη εγκληματικότητα να μην εισχωρήσει. Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει. Να προσθέσω κι εγώ κάτι που νομίζω σχετίζεται με αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Στην τρίτη διαφάνεια περί αμοιβαία αναγνώρισης είπατε πω το Συμβούλιο, το δικαστήριο με θεωρούσε πως ε, η παροχή η μη σύνομη παροχή παιχνίων σε άλλη χώρα σημαίνει πως ε, δεν, δεν μπορεί να υπάρχει διασφάλιση προστασίας των καταναλωτών. Αποκλείεται έτσι κάποια πανευρωπαϊκή αδειοδότηση ε, με τρόπο που θα υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή εφαρμογή. Βεβαίω κάτι τέτοιο θα έπρεπε να το κάνει η Κομισιόν. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ πρακτικό, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα με βάση την εκτεταμένη νομολογία. Άλλα σχόλια. Ωραία, θα δώσω τον λόγο άρα στους ε, ομιλητές μας για να απαντήσουν σε αυτά τα σημεία. Για να απαντήσω σε αυτά. Είναι πάρα πολύ καλό το σχόλιο αυτό με τους ορισμούς. 85% των site χωρίς άδεια. Ε, δεν έχω δει στατιστικά στοιχεία αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην Ευρώπη και μετά υπάρχει το πρόβλημα του ορισμού εντός της Ευρώπης του τι είναι ισχύουσα άδεια σε ένα κράτος μέλος και σε ένα άλλο. Για το θέμα των συμμαχιών, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως όταν ρυθμίζουν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να επανεφεύρουν τον τροχό, οπότε υπάρχουν κάποιες συμμαχίες, παραδείγματο χάρη καταλαβαίνω πως η Δανία συζητάει με μια υπεράκτια δικαιοδοσία έτσι ώστε η τεχνική υποδομή να επιτραπεί στην Δανία και βλέπουμε πως η Γαλλία και η Ιταλία θα υπογράψουν διμερή συμφωνία αργότερα εντός του μηνός. Ε, δεν είναι μόνο από ρυθμιστική σκοπιά οι τεχνικές σκοπιές που πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά και από την εμπορική σκοπιά. Βλέπετε πως η ανάγκη για κάποιες ε, συμμαχίες ε, π.χ. κρατών μελών ε, μικρών, όπως η Δανία με μικρό αριθμό παικτών, για να υπάρξει μια ελκυστική ρυθμισμένη από τις αρχές προσφορά, σημαίνει πως θα υπάρχει κάποια ρευστότητα για αυτά τα παιχνίδια ζητήματα τα οποία βεβαίως δεν έχει να αντιμετωπίσει παραδείγματος χάρη η Ιταλία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συμμαχίες, περισσότερο ως απόρρια πρακτικών ζητημάτων για να ε, λειτουργήσει η αγορά. Όχι από καθαρά νομική σκοπιά, αλλά ε, υπάρχουν κάποιες, κάποιες συμμαχίες που παρακολουθούμε εμείς και για αυτό το οποίο είπατε για την αμοιβή αναγνώριση. Υπάρχει ε, αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και ξέρω πως ε, συζητάνε οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ε, τα του τζόγου. Οπότε νομίζω πως θα μπορούσαν να βρουν μια λύση μέσω των συναντήσεων γκρεφ κτλ. Ευχαριστώ. Κύριος Φλέμινγκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μπαίνουμε στην καρδιά της ε, συζήτησης. Αν είχαμε λίγες εβδομάδες, ε, ευχαρίστω να συνεχίσω, αλλά νομίζω αυτό επαφίεται στο Κοινοβούλιο. Ε, Επίτρεψατε μου να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε το δικαστήριο στην παράγραφο 130 σε μία από τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του, όπου λέει Προκύπτει άρα πως κάθε κράτος μέλος ε, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, να προσφέρει τη γερά παίγνια εντός της επικράτειάς του, να έχει άδεια που έχει εκδοθεί από τις δικές του αρμόδιες αρχές, ανεξαρτήτως του εάν έχει άδεια εκδοθεί σε άλλο κράτος ε, μέλος. Οπότε το δικαστήριο κατέστησε σαφές πως ε, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των τυχερών παιγνίων δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι μια απλή οικονομική δραστηριότητα και θυμάμαι μάλιστα πως υπήρχε συζήτηση για το εάν είναι καν οικονομική δραστηριότητα και άρα είναι εντό αρμοδιότητας του ΔΕΚ το δικαστήριο έκρινε πως είναι οικονομική δραστηριότητα αλλά με ιδιαίτερη φύση και ε, δεν μπορούν έτσι να ισχύσουν ε, απλά όλοι οι κανόνες. Π.χ. δεν μπορούν ε, να ισχύσουν έτσι απλά οι κανόνες του ανταγωνισμού και μίλησε για οικονομικές, πολιτικές ε, και κοινωνικές διαφορές που δείχνουν κατά την άποψή μου το πόσο πλούσια είναι η Ευρώπη από χώρα σε χώρα και άρα μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν διαφορετική άποψη για το πώς θα ρυθμίσουν την αγορά του τζόγου. Και αν δείτε την αγορά του τζόγου στη Φιλανδία είναι διαφορετική από αυτή στην Ιταλία ή ε, στην Ελλάδα. Και Νομίζω πως βασίζεται σε συγκεκριμένες αξιολογήσεις και επιλογές πολιτικές που έχουν γίνει και το επέβαλε αυτό, το επανέλαβε το 1999 το δικαστήριο λέγοντας πως ανεξάρτητος ήταν τα άλλα κράτη-μέλη, το κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει τον τύπο των παιχνιδιών, τον όγκο των παιχνιδιών, το πώς θα γίνει μέσω μονοπωλίου ή μέσω μιας άδεια κτλ. Οπότε όλα είναι δυνατά στην Ευρώπη, εξαρτάται λοιπόν από τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, δηλαδή Κομισιό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Αν αυτά τα θεσμικά όργανα μπορούν να βρουν έναν τρόπο να πούν θέμε μια πανευρωπαϊκή άδεια, τότε τελείωσε. Αλλά έχοντας ε, εξετάσει το τι λένε τα κράτη-μέλη στο δικαστήριο και το τι συζητάνε στο Συμβούλιο, απέχουμε πολύ από μια τέτοια λύση. Οπότε όταν λέω πως απαιτείται μια πολιτική λύση, δεν νομίζω πως μπορούμε να περιμένουμε ένα όνειρο μία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στο τζόγο, ακόμη και αν θέλαμε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε πως οι λύσεις αυτές προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Η πολιτική λύση είναι αναγκαία, γιατί βλέπουμε σε όλα τα κράτη-μέλη πάρα πολλές υποθέσεις που πάνε στα δικαστήρια και δημιουργούν αστάθεια. Γι' αυτό απαιτείται μια πολιτική λύση. Το δικαστήριο έχει πει ξανά και ξανά ως έχει το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο αυτή τη στιγμή. Ε, ξεκάθαρα δηλαδή λέει πως ε, έτσι έχει συνθήκη και δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Οπότε επαφίεται στον νομοθέτη. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να βρεθεί μια λύση με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητα. Αυτό δεν σημαίνει πώ δεν μπορεί να κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη. Απαιτείται μια διτή προσέγγιση όπου αποφασίζουν για το περιβάλλον τα κράτη-μέλη και ε, μπορούν να υπάρχουν περαιτέρω κανάνες, π.χ. ακαιρεότητα του αθλητισμού, διαφημίσεις, κοινό αγώνας κατά της εξάρτησης, της απάτης, π.χ. δεν είναι λογικό κάποιος εξαρτημένος να αποκλείεται σε ένα κράτος μέλος, αλλά να μπορεί να τζογάρει σε άλλο κράτος μέλος. Τέτοιου κανόνες θέμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτοί οι κανόνες μπορούν να δημιουργήσουν σταθερότητα. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αυτά που είπατε βρίσκονται στον πυρήνα του ζητήματο, που θα ακολουθήσουν την έκθεση του κυρίου Κρόιτσμαν και την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής, αλλά τώρα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με συναφή ζητήματα, πώς ε, λειτουργούν οι ρυθμιστικέ αρχές, κάποια οικονομικά, κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα καταναλωτών. Αυτά θα μα απασχολήσουν στα δύο επόμενα τμήματα της συζήτησή μα. Έχουμε τέσσερι ομιλητέ. Πέντε λεπτά έχετε εκαστός, θα σας και εσάς. Ζων Φρανσουά Βιλότε, που είναι πρόεδρος ε, της ε, της Γαλλικής ε, ρυθμιστική αρχή για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση, Αγζέλ ονομάζεται, ο Δόκτωρ και Φράνσε, που έρχεται από την καγκελαρία του Ομόσπονδου Κρατηδίου Σάξονι Ανχάλτ από τη Γερμανία, ε, κατόπιν ε, ε, θα δούμε τα θέματα των στοιχημάτων, γιατί υπάρχουν ε, γερμανικά ζητήματα, κάποια ομοσπονδιακού χαρακτήρα ζητήματα, θα μα τα πείτε εσεί, Πίτερ Ρέινολ στη συνέχεια, που εκπροσωπεί την Ένωση για την εξαποστήριξη για τα εξαποστάσεως τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα και κατόπιν Φρίτριχ Στίκλερ από τις Ευρωπαϊκές ελαχιοφόρους Αγορές, είναι πρόεδρος της οργάνωσης European Lotteries. Θα σχολιάσει το θέμα των λαχείων και λαχιοφόρων αγορών. Αρχίζουμε με τον Ζαν Φρανσουά Βιλότ, πέντε λεπτά. Έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός. Θα κάνω απολογισμό των όρων ε, ανοίγματο τη αγορά για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση στη Γαλλία. Η Γαλλία τροποποίησε την νομοθεσία τη ε, το Μάιο του 2010 βάσει μιας διπλής διαπίστωσης. Πρώτον, ότι δεν υπήρχε κάποια δυνατή αυτορύθμιση. Αν δεν υπήρχε δηλαδή ισχυρή δημόσια ρύθμιση, δεν εξασφαλίζαμε τέσσερι βασικούς στόχους. Καταπολέμηση των εθισμών, προστασία των ανηλίκων, ε, καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, ε, νομιμότητα των δραστηριοτήτων ε, σε απευθεία σύνδεση, κυρίως όταν μιλάμε για δικτυακούς τόπους προσφέρουν στοιχήματα και κατόπιν ισορροπία στην ίδια την αγορά. Εάν δεν υπάρχει δημόσια ρύθμιση, ελοχεύουν συστημική υψηλή κίνδυνη, μπορεί να απολέσει πάσα αξιοπιστία το σύστημα και η αγορά μπορεί και να εκλείψει εάν δεν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της δεύτερη διαπίστωση, η ιδιαιτερότητα των ε, ε, παιχνιδιών σε απευθεία σύνδεση. Αυτό είναι το παράδοξο του μονοπωλίου και της ε, ποσοτικής ρύθμισης. Όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε μια εσωτερική αγορά και αν δεν προσφέρεται σε σχέση με αυτή τη ζήτηση μια αρχή μονοπωλίου, τότε αυτή η ζήτηση θα προσανατολιστεί προς την παράνομη προσφορά που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να καταπολεμήσει γκρεμίσει κανείς ε, στο διαδίκτυο. Ε, όταν λοιπόν το μονοπόλιο προσφέρει με ε, περισσότερες υπηρεσίες για να καλύψει τη ζήτηση, τότε διατρέχει κινδύνους ενώπιον της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Επιτίθεται ζήτημα νομιμότητας. Οπότε η Γαλλία άνοιξε την αγορά των τυχερών παιχνιδιών σε τρία μονοτμήματα. Τυχερά παιχνίδια ε, όπου χρειάζεται κάποια δεξιότητα από πλευρά του παίκτη, τα στοιχήματα για τι υποδρομίε και το πόκερ. Ε, οι αδειοδοτήσει χωρούνται βάσει μια ε, προσφορά με ποσοτικά στοιχεία, ώστε να κατοχυρωθεί η διαφάνεια για τα κεφάλαια του φορέα εκμετάλλευση, καθώ και η όλη διαδικασία, δηλαδή τα λογισμικά παιχνιδιού που χρησιμοποιούνται, αν είναι ασφαλή, παραδείγματο χάρη. Και τρίτον, οι φορείς εκμετάλλευση έχουν ε, την υποχρέωση να έχουν ε, συστήματα πληροφορικής ε, στη Γαλλία τέτοια ώστε η ρυθμιστική αρχή να έχει πρόσβαση στο σύνολο των συναλλαγών ανάμεσα στους εγκεκριμένου καταχωρημένους φορείς εκμετάλλευση και τους παίκτες. Δεν υπάρχει περιοριστικός αριθμός αδειών, δεν υπάρχει όριο φορολογικό στη Γαλλία, υπάρχει μόνο η αποχρέωση απόλυτης διαφάνειας και απόλυτης ανιχνευσιμότητας απολογισμό τώρα ε, για τον ένα χρόνο ε, λειτουργία. 500 ε, άδειε έχουν εκδοθεί 35, ε, από 35 διαφορετικέ επιχειρήσει που έχουν την έδρα του ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 δι ευρώ στοιχημάτων περίπου που κατέγραψαν οι εγκεκριμένοι φορεί εκμετάλλευση. Τα ποσά αυτά κυρίω βρίσκονται στου φορεί του πόκερ και των παιχνιδιών μετρητών 500 ε, εκατομμύρια για αθλητικά στοιχήματα και 800 έως 900 εκατομμύρια για τα ε, ε, στοιχήματα υποδρομίας. Τα spread betting, τα στοιχήματα για τα spread απαγορεύονται και τα επικά στοιχήματα ισχύουν μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυξήθηκε πάρα πολύ διαφάνεια στην αγορά τον τελευταίο χρόνο. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους επιγραμμικούς παίκτες. Έγιναν διάφορες στατιστικές μελέτες από τη διοικητική ε, αρχή της οργάνωσής μας, οργάνωση όπου προεδρεύω. Χάρη σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία ξέρουμε ποια είναι η ηλικία, αν είναι ενήλικες οι παίκτες, ε, το φύλλο τους, ε, πώς, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν, πού συγκεντρώνουν τα περισσότερα στοιχήματά τους. 10% των παίκτων εκπροσωπούν 83% των στοιχημάτων, 15% αντιστοιχημάτων στοιχεί στο 50% των στοιχημάτων. 15% των παικτών, 50% των στοιχημάτων. Βλέπετε το πρόβλημα τη παρακολούθηση των τυχερών παιχνιδιών. Το θέμα του εθισμού δεν είναι ένα θεωρητικό πρόβλημα. Ε, επίσης ε, αυτόματοι συντονιστές των παιχνιδιών ε, που υποχρεωτικά υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι. Οι ανήλικοι δεν μπορούν φυσικά να παίξουν. Οι φορείς εκμετάλλευσης οπωσδήποτε πρέπει να έχουν εξουσιοδοτημένα λογισμικά και οι φορείς των στοιχημάτων υπακούν σε πάρα πολύ αυστηρούς όρους. Δεν μπορούμε να στοιχηματίσουμε όσα λεφτά θέλουμε οπουδήποτε και οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει σχέση ανάμεσα για τη, διοργανωτέ των αθλητικών ε, εκδηλώσεων, αθλητικών συναντήσεων και του φορέα εκμετάλλευση που προσφέρει στοιχήματα για αυτή τη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση. Εδώ και ένα χρόνο, για να κλείσω σιγά σιγά, παρατηρούμε ότι είναι αποτελεσματική η εθνική ρύθμιση τη αγορά και ενώ υπήρχε ε, επιγραμμικώ ε, παράνομη προσφορά τυχερών παιχνιδιών σε ποσοστό 80 με 90%, σήμερα έχουμε φτάσει σε νόμιμη προσφορά στα ίδια επίπεδα. 80 με 90% τη προσφορά παιχνιδιών στη Γαλλία. Δεύτερον, προφανώς υπάρχει περιθώριο για να ρυθμίσουμε καλύτερα κάποια ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο θα αναφέρω. Ε, καταπολέμηση κατά πολέμηση των παρανόμων δικτυακών τόπων ε, είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν τόσο ώστε ε, να υπάρξει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία τους. Δεύτερη διαπίστευση γιατί το ήθος, το αθλητικό ήθος δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι παρά την εθνική προστασία προστατεύουμε ε, το άθλημα ε, σε σχέση με τα στοιχήματα της εγχώριας αγοράς αλλά και της ε, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, thank you very much uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική σας τα όσα μας αναφέρετε περί σίγουρα θα σας θέσουμε και ερωτήσεις ε, για όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ο Δόκτωρ Φραντς. Ευχαριστώ. Χαίρομαι μπορώ να μιλήσω σήμερα ενώπιον σας. Μία ρύθμιση των τυχερών παιγνίων δεδομένων των πάρα πολλών πολιτισμικών και κοινωνικών παραδόσεων και των στάσεων των κρατών μελών μπορεί να γίνει μόνο σε εθνικό επίπεδο. Διαφορετικά ρυθμιστικά μοντέλα υπάρχουν μέσω των οποίων θα πρέπει να επιλέξει ο εθνικός νομοθέτης εάν θα πάμε σε απαγόρευση ή μη, εάν θα υπάρχει αυστηρή αδειοδότηση μέχρι ε, πλήρης απελευθέρωση. Στην ε, Γερμανία υπάρχει στόχος του νομοθέτη που είναι προστασία της κοινωνίας και του παίκτη. Αυτό οδηγεί μεταξύ άλλων σε αυστηρές απαιτήσεις για την διαμόρφωση του τι προσφέρεται στο διαδίκτυο. Τα γερμανικά κρατήδια έχουν συνάψει μία σύμβαση ε, που ετέθη ενισχύει από 1η Πρώτου 2009 και 31 Δωδεκάτου ε, του 11 λίγη και άρα θα πρέπει να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία η διάσκεψη των αρμοδίων υπουργών των κρατηδίων. Σχέδιο νέας σύμβασης έχει ήδη δοθεί τον Απρίλιο του 2011 στην ε, Κομισιόν. Τι γίνεται τώρα με το διαδίκτυο. Η απαγόρευση βεβαίως υπάρχει για να μειωθεί η εξάρτηση και άρα καταρχήν η προσφορά και να αξιθεί το κατόφλι συμμετοχή και έχει επιβεβαιωθεί και από το δικαστήριο το συνταγματικό το γερμανικό και το ΔΕΚ. Ο στόχος ο οποίος υπάρχει τώρα δηλαδή να διασφαλιστεί μία κάποια προσφορά και να παραμείνει εντός νομίμων πλωσίων η ανάγκη του πληθυσμού ε, θεωρούμε πως ε, δεν έχει καλυφθεί από τη σύμβαση που έχουν υπογράψει μεταξύ του στα κρατήρια και αυτό επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων από τη μεγάλη παράνομη προσφορά που υπάρχει στο δίκτυο. Υπήρχε λοιπόν μια ανάλυση που υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2009 και έγινε κατόπιν παραγγελία των ε, κρατηδίων και βλέπουμε πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, εξάρτησης, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε ειδικά για παιχνίδια στοιχήματος ε, στον, σε αθλητικά γεγονότα και καζίνο. Από ό,τι φαίνεται όμως πως η πλήρης απαγόρευση αποτελεί ένα στόχο ο οποίος δεν θα επιτευχθεί. Θα υπάρχουν πάντα κάποιοι οποίοι θα προσφέρουν και κάποιοι οποίοι θα τζογάρουν. Οπότε η ανάλυση λέει στην περίπτωση η οποία, στην οποία δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος στο διαδίκτυο θα πρέπει να υπάρχει μια διοδότηση περιοριστική υποκρατικό έλεγχο. Τώρα, ποια είναι η πρόταση της νέας αυτής συνθήκης ε, περί τυχερών παιγνίων η οποία έχει κοινοποιηθεί στην ε, Κομισιόν. προβλέπεται πρώτα απ' όλα η αδειοδότηση για όσους ε, σκοπεύουν να σχηματίσουν σε καζίνο, σε πραγματικά παιχνίδια και στο διαδίκτυο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ε, να δοθεί μια εναλλακτική η οποία θα είναι νόμιμη και θα προστατεύει την ε, νεολαία και τυχόν εξαρτημένους. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες αλλαγής που έχει το διαδίκτυο και εδώ πέρα σημαίνει πως δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, είναι πάρα πολύ εύκολο και άνετο να παίξει κανεί. Επίσης υπάρχει ένα εφέ σύμφωνα με το οποίο δεν αντιλαμβάνεται πλέον κανείς κάτι το, ως κάτι το επικίνδυνο κάτι το οποίο κάνει στο διαδίκτυο και βεβαίως ο ιδιαίτερος κίνδυνος που διατρέχουν είναι νεαροί παίκτες. Οπότε, για το στοίχημα online και τις ε, λοταρίες ε, online ε, προβλέπεται εάν τηρηθούν αυτοί οι όροι να επιτραπεί κάτι τέτοιο στο διαδίκτυο. Το αντίθετο ισχύει για τα καζίνο γιατί θεωρείται πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος και καταλήγουν η συμμετοχή Ε, σε ε, ένα ψηφιακό καζίνο θεωρείται ότι δημιουργεί λιγότερη εξάρτηση από ότι ε, σε ένα πραγματικό. Άρα θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη ρύθμιση αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Σας ευχαριστούμε που τήρησατε και το χρόνο και εσείς. Να περάσουμε στον κύριο Πίτερ Ρέινολτς από την Ένωση Τυχερών Παιχνιδιών Εξ Αποστάσεων. Έχετε κάποιες διαφάνειες νομίζω, ναι. Έχω κάποιες διαφάνειες, θα τις δείτε στην οθόνη. Να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εκπροσωπώ λοιπόν εδώ την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Παιχνίων και Στοιχημάτων ε, ε, και την Ένωση Τυχερών Παιχνιδιών Εξαποστάσεων προτεκτελεί έναν από τους ορθισμένους κλάδους στην Ευρώπη. Είμαστε επικεφαλής στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και προσφέρουμε καινοτόμα και ασφαλή παιχνίδια. Θεωρούμε ότι η Πράσινη Βίβλος αποτελεί μια ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά και ελπίζουμε ότι θα είναι το πρώτο βήμα προς να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να απαντά στην πραγματικότητα της αγοράς ε, γιατί ε, ο, τα τυχερά παιχνίδια εξαποστάσεως είναι εδώ και είναι εδώ για να μείνουν. Αν ε, χάσουμε την ευκαιρία τότε δεν θα μπορέσουμε ούτε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές ε, και τη δημόσια τάξη και βλέπουμε ότι τα τυχερά παιχνίδια, τα επιγραμμικά αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα του ηλεκτρονικού εμπορίου ήδη. το πολιτική ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι σημαντική ε, σε αυτό το πλαίσιο έτσι λοιπόν, να σας ε, δώσω εδώ το ιστορικό σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς. Όπως βλέπετε, έχουμε μια τεράστια ίδια αγορά. Μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια εσόδων ε, το 2010 και η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου εκπροσωπεί το ίμιση ε, των παγκόσμιων επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών. Βλέπετε ότι μιλάμε εδώ για 11% μόνο το 2010 για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μερίδιο της αγοράς, ε, ο παραδοσιακό μοντέλο εξ αποστάσεως θα συνεχίζει να έχει το, τερά, το μερίδιο του λέοντος, ε, όμως βλέπουμε ότι πρόσθετα ε, ε, έσοδα ε, προέρχονται από τον επιγραμμικό τομέα. Το βλέπουμε αυτό και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Βέβαια έχουμε και τις λαχιοφόρους αγορές που είναι σε μονοπωλιακή λειτουργία Επίσης ε, βλέπουμε ότι έχουμε και δευτερεύουσες ε, επιχειρήσεις όπου επωφελούνται από τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια όπως είναι η διαφήμιση, η χρηματοοικονομικά κτλ. Ε, τα τυχερά παιχνίδια υπόκειται σε ε, αυστηρή νομοθεσία όσο και περισσότερα κράτη-μέλη προσπαθούν ε, να ρυθμίσουν τον κλάδο. Η συζήτηση σήμερα είναι ότι θα έχουμε πρόσβαση σε σωστά ρυθμισμένες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες και ακολουθήσαμε κοινή κίνδυνη να μην προσφέρουμε ανταγωνιστικές προσφορές γιατί θα υπάρχει πρόσβαση των παικτών στη μαύρη αγορά. Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόσβαση πρόβλημα ε, δεν ε, συνάδει η σημερινή κατάσταση με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα τομέα που είναι διασυνοριακός εκφύσεως ε, το να έχουμε 27 αριθμιστικά μοντέλα δεν είναι κάτι που επιθυμεί κανείς χρειαζόμαστε μια σειρά κοινών προτείνων για να θέσουμε το πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα καλύψαμε ήδη. Ότι είχαμε πάρα πολλέ υποθέσει ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχει μεγάλη ε, αβεβαιότητα δικαίου. Τα πράγματα δεν μπορούν να παραμείνουν ω έχουν. Ε, σε αυτού του οικονομικού καιρού είναι ζωτικό η Κομισιόν να διαδραματίσει το ρόλο τη ώστε με το φύλακα τη συνθήκη και να προστατεύσει τι αρχέ που περιλαμβάνονται στη συνθήκη και να αποτρέψει τον περαιτέρω κατακαιρματισμό τη εσωτερική αγορά. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ, λαϊχοφόρη αγορά, ρυθμιστέ, ε, κυβερνήσει, επιχειρήσει, όλοι μα είμαστε δεσμένοι σε υπεύθυνα τυχερά παιχνίδια. Ε, υπάρχουν μηχανισμοί για την άμβληση τη κοινωνική ζημία. Υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Ο κλάδο μα είναι ήδη ψηλά ρυθμισμένο. Πρέπει να σεβόμαστε τι απαιτήσει ε, άδεια, να προστατεύουμε τα δεδομένα να σεβόμαστε την εταιρική νομοθεσία, να σεβόμαστε την νομοθεσία για ε, την ομοποίηση παράνομων εισόδων και επίσης ε, επιλέγουμε και εμείς ε, κάποια νομοθεσία για να αυξήσουμε τα πρότυπα ή προστασία του καταναλωτή, κυρίως των ανηλίκων και των ευπαθών καταναλωτών. Κάτι τέτοιο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία. Ο μόνος λόγος που ένας καταναλωτής θα σκεφτόταν μόνο να πάει στην παράνομη πλευρά κρατώντας την πιστοτική κάρτα είναι επειδή η ρυθμισμένη αγορά έχει απαντήσει στη ζήτηση που υπάρχει για την προστασία των παικτών και στην προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Ω ε, κλάδος εμεί προσπαθούμε να πάμε και παραπέρα μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μαζί με τη ΣΕΝ ε, έχουμε αναπτύξει 134 συγκεκριμένα μέτρα που διασφαλίζουν ε, τι θεμητέ πρακτικέ για τα τυχερά παιχνίδια και προστατεύουν του καταναλωτέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα building block για πανευρωπαϊκά πρότυπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ε, που τηρήσατε το χρόνο και τώρα σε αυτό το τμήμα έχουμε τον κύριο Στίκλερ ο οποίος είναι πρόεδρος ε, των Ευρωπαϊκών Λαχυροφόρων Αγορών και αυτός έχει κάποιες διαφάνειες και νομίζω μας έχει στείλει και ένα έγγραφο. Νομίζω ότι το έγγραφό σας θα, για να το παρουσιάσετε θα χρειαστεί παραπάνω από πέντε λεπτά. Ναι, ευχαριστώ. Σας, δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που προσκαλέσατε τις ε, ευρωπαϊκές λοταρίες. Ε, να σας δώσω, να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του οργανισμού μας. Είναι ένα σύνδεσμος κρατικών ε, λοταριών και κυρίως μιλάμε βεβαίω σε προγνωστικά αθλητικά για κοινωνικό όφελος. Ναι, αυτή είναι η διαφάνεια. Είμαστε λοιπόν η μόνη ένωση με μέλη και από τα 27 κράτη-μέλη. Όλα μας ε, τα μέλη προσφέρουν παιχνίδια ε, με ε, άδειε στις επικράτειες αυτές και σέβονται εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Δεν πουλάμε διασυνοριακά. Το 2010 συνεισέφεραν τα μέλη μας γύρω στο... 25 δισεκατομμύρια ευρώ στους κρατικούς προϋπολογισμούς και σε καλούς σκοπούς όπως π.χ. πρόθεση αθλητισμού, πολιτισμού κτλ. Οπότε μιλάμε για ένα κοινωνικό μοντέλο. Μου ζητήθηκε σήμερα να εξηγήσω την άποψή μας για το πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθεί σε αποτελεσματική ρυθμίση και έλεγχο του τζόγου στο διαδίκτυο. Εδώ πέρα θα ήθελα να πω Πάμε παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Πώς ε, πριν από δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εθέτησε το πρώτο του σχετικό ψήφισμα με βάση την έκθεση Μόζε και εμείς ε, συμφωνούμε πλήρως με το περιεχόμενο του ψηφίσματος εκείνου και προτείνουμε το επερχόμενο ψήφισμα του Κοινοβουλίου να βασιστεί στο προηγούμενο. Το ψήφισμα του 2009 εγκρίθηκε με πλειοψηφία 85% και ε, κοιτάζοντας σχεδόν 40 παρεμβάσεις που έκαναν στη συζήτηση της Ολομέλειας ε, οι Ευρωβουλευτές, χαιρόμαστε για το ότι αυτή η θέση ε, βρίσκει τη στήριξη και του Κοινοβουλίου σε αυτή τη θητεία. Η μεγαλύτερο πλεονέκτημα της έκθεσης Σαλτεμόζε είναι πώς ορίζει τις βασικές, τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αλληλεγγύη, ακαιρεότητα, επικουρικότητα και προφύλαξη. Το μοντέλο του δημοσίου ωφέλους που καθοδηγείται με βάση αυτές τις αρχές έχει αποδειχτεί το καλύτερο μοντέλο εδώ και πολλές δεκαετίες. Επειδή βεβαίως η πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί στην ε, τεχνολογική αλλαγή, δεν θα ήταν σωστό να ξεχάσουμε αυτές τις αρχές, ειδικά όταν υπάρχει τόσο ευρεία συνένεση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών, όχι μόνο εδώ μέσα, αλλά και στο Συμβούλιο και στο ΔΕΚ. Οπότε, έχω και λίγο χρόνο, θα ήθελα ε, να μην αναφέρω πολλά πράγματα. Έχετε τις 8 σελίδες που σας έχω μοιράσει, αν θέλετε ρίξτε μια ματιά. Να πω μόνο κάποια πράγματα για την αρχή της ακεραιότητας. Ήδη το 10 έχει ξεκαθαρίσει πολλά σημαντικά νομικά ζητήματα. Δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, πρέπει να υπάρχει εθνική άδεια κτλ. από την υιοθέτηση της έκθεσης Σαλτεμόζε. Το επόμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει και μπορεί να πάει πολύ παραπέρα γένεια της ακεραιότητας πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την πλήρη συμμόρφωση και την αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας. Είναι μια ε, συχνή παρεξήγηση πως η παράνομη παροχή τέτοιων υπηρεσιών διασυνοριακά ε, στο ίντερνετ προέρχεται ε, εκτός Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι εντός της Ευρώπης, εξού και η ανάγκη ευρωπαϊκής δράσης για να λύσουμε το πρόβλημα. Ε, για να εξηγηθώ, η Γαλλία η οποία όπως ακούσαμε μέρη άνοιξε την αγορά αυτή πέρσι, οι ρυθμιστικές αρχές έστειλαν εκατοντάδες προειδοποιήσει ε, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο που δεν έχουν άδεια γαλλική αλλά προσφέρουν υπηρεσίες στη Γαλλία. 80% των εταιριών αυτών ε, βρίσκονται εντό τη Ένωση. Αλλά να έρθει το σημαντικότερο για εμένα. Για λόγου προστασία των καταναλωτών και δημόσια τάξη, αλλά και για να υπάρχει χρηματοδότηση ε, σκοπών δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει οι κατέχοντες εθνικής ε, εθνική άδεια να προστατευτούν από παράνομο τέτοιο ανταγωνισμό. Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά από μόνες τους ε, διασυνοριακές συναλλαγές. Εδώ πέρα χρειάζεται σε συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να έχουμε κάποιες ρυθμιστικές αρχές με βάση τις οποίες και εδώ πέρα συνιστώ αυτό το μοντέλο μία εταιρεία θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί ή να υποβάλει προσφορά για εθνική άδεια εάν μπορεί να αποδείξει πως δεν λειτουργεί αντίθετα με τον νόμο σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι διαφορετικές απόψεις που ακούμε. Έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Αλλά πρωτού περάσουμε σε αυτό το τμήμα, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών ε, της κυρίας Γκέπχαρντ που εργάζεται άοκνα στην Επιτροπή μας. Ε, ε, ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε θέσεις για όλους, διότι σήμερα υπάρχει αυτή η ακρόαση, αλλά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν. Α περάσουμε σε ένα γύρο ερώτα απαντήσεων. Ο κύριος Φόξ μου ζήτησε πρώτος το λόγο, οπότε παρακαλώ μετά ο εισηγητής, ο κύριος Κρόιτσμεν, ο κύριος Άμπατ, ποιος άλλος, κυρία Γκέπχαρτ. Και ο κύριος Κόχολα μετά από όλους αυτούς. Ο κύριος Φόξ αρχίζει. Ε, προς τον Δόκτωρ Φρανς ε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Το 2008 ε, η Φόρσα, ε, ερευνητικό ίδρυμα της Γερμανίας, ε, ανέφερε ότι 2,2 εκατομμύρια τακτικά παίζουν στο διαδίκτυο παρότι ουσιαστικά είναι παράνομο. Αυτό σε συνδυασμό με τα 4 εκατομμύρια παικτών όπου είναι νόμιμα αυτά τα παιχνίδια και ρυθμισμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε η απαγόρευση δεν, έχει, δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Τι πιστεύετε, δεν είναι καλύτερο να ρυθμιστεί αυτή η αγορά και έτσι να να προστατευτούν οι καταναλωτές παρά να αγνοούμε την αγορά και να επιβάλλουμε απαγόρευση που αγνοείται τελικά από όλους και είναι ε, επιβλαβής για τους καταναλωτές. Κύριε Κρόιτσμαν, έχετε άλλη ερώτηση ή θέλετε να τοποθετηθείτε γι' αυτό μήπως? Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Φόξ. Ε, θα μιλήσω γερμανικά. Είδαμε το, το φάσμα Είδατε από τη Γαλλία που το έχει ρυθμίσει. Έχουμε τα παράνομα στοιχήματα. 80 90% γίνανε πλέον νόμιμα και ο κύριος Στίκλερ είπε πως ε, να διατηρηθεί το μονοπόλιο, δηλαδή να μην έχουμε online διασυνοριακό στοίχημα. Και είναι ζήτημα επιβολής, να τηρηθούν οι κανόνες. Κάτι το οποίο οπωσδήποτε ε, θέλει να κάνει και η γαλλική πλευρά. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα προς ε, την κυρία Φραντς. Τα κρατήδια τα γερμανικά προσπαθούν να βρουν ένα νέο τρόπο και να πούνε πως θα ανοίξουμε λίγο την αγορά αλλά μόνο για 6-7 εταιρείε. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ε, χώρες όπως ε, κρατήδια όπως το Σλέσφιχ Χόλστάιν έχουν κάνει δική τους πρόταση και θέλουν να διατηρήσουν το μονοπόλιο αλλά να έχουν ε, και να μην διατηρήσουν το μονοπόλιο αλλά να έχουν μια ελεύθερη αγορά η οποία θα έχει άδειε. Γιατί ε, όπως σας είπα οι δικές μου οι είναι αυτές και άρα όλες οι εταιρείες θα μεταφέρουν την έδρα τους στο Σλέσβι Χόλσταν και από εκεί πέρα θα πάρουν άδεια. Ε, τι θέλετε, πώς σκοπεύετε λοιπόν ε, να περιοριστείτε σε 7-8 εταιρεία όταν μόνο στη Μάλτα υπάρχουν εκατοντάδε. Χωρί να έρθετε μετά σε σύγκρουση με το δικαστήριο. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι είστε ο πιο δημοφιλής, Dr. Franz. Όλοι σας απευθύνουν ερωτήσεις. Βέβαια μπορεί να αλλάξει αυτό. Ο κύριος Άμπατ. Ευχαριστώ. Για να αλλάξουμε και λίγο θα θέσω ερωτήσεις εγώ στους, ε, στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Σε σχέση με αυτό που μας είπε ο κύριος Βίλωτ και ο κύριος Τίνλερ για το θέμα της ισορροπίας ε, στις αγορές ως προς τη χρηματοδότηση και αυτό που μας είπε για την ε, ακαιρεότητα, το ήθος στις αθλητικές εκδηλώσεις και για τα στοιχήματα. Ακούσαμε κάποιες για την οδηγία σχετικά με την προστασία των βάσεων δεδομένων. Ποιε είναι οι αρχές που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν την αγορά των στοιχημάτων και εφόσον θέλουμε να προαγάγουμε το ήθος ε, στον αθλητισμό και θέλουμε να πλαισιώσουμε τα αθλητικά στοιχήματα, Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Θα προσφέρει μια επαρκή νομική βάση αυτή η οδηγία για να μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Και τέλο, ε, για την οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο ε, βρώμικου χρήματο. θα μπορούσαμε ενδεχομένω να εξετάσουμε την ενδεχόμενα επέκταση στο πεδίο εφαρμογή για να καλυφθεί ο τομέα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κέπχαρτ. Äh, πάρα πολύ θα ήθελα να αναφερθώ ακόμη μια φορά στο θέμα της ε, χρηματοδότησης ε, και των ε, κερδών, το οποίο δεν ανέφερε κανένας ομιλητής. Και κάτι το οποίο έχει σημασία για τη ρύθμιση γενικότερα και για τους ανθρώπους που αποτελεί το κίνητρο για να παίξουν τυχερά παιχνίδια και το πώς έχει ρύθμιση στα διάφορα κατημέλη. Εκεί βεβαίως που υπάρχει απαγόρευση δεν υπάρχει αναδιανομή των κερδών αυτών, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω εκεί όπου υπάρχουν άδειες ε, πόσο, πιο ποσοστό των χρημάτων αναδιανέμεται και πού πάνε τα λεφτά που δεν ε, διανέμονται μετά. Και αυτό με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Κόπουλα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, στον κύριο Κρότσμαν, γενική ερώτηση. Γιατί οι εταιρείε, ε, οι ρυθμιστικές αρχές δεν εφαρμόσουν τεχνικές λύσεις ε, για να αποφευχθεί η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα οποιονδήποτε κατάχρησης, ξεπλήματος, βρώμικου χρήματος κτλ. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αποφευθούν αυτοί οι περιορισμοί με διάφορα τεχνάσματα. Αν αναφερθείτε, το χάρη, στις γενικές προϋποθέσεις χρήστη. Και μια ακόμη ερώτηση σε σχέση με την ταυτοποίηση του παίκτη. Να τη θέσω στον κύριο Βιλότ. Η ταυτοποίηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρχικό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν ε, τέτοια τυχερά παιχνίδια χωρίς να υπάρχουν όρια παρακολούθηση, ε, γιατί επιτρέπετε κάτι τέτοιο, ποια είναι η άποψή σα ε, στο να δημιουργηθούν όρια, να τεθούν κάποια όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν εξετάζουμε το θέμα της στήρησης χρημάτων σε διαφορούς λογαριασμούς. Κάτι τέτοιο διευκολύνει την, την νομιμοποίηση παρανομών εισόδων. Και διευκολύνει να κινούνται τα χρήματα χωρίς να υπάρχει πρόσβαση ε, των ελεκτικών αρχών και των φορολογικών αρχών. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ε, Τις ε, πρώτες ερωτήσει, ε, τις απευθύνεται στον κύριο Ρέινολτς ε, και αν και αναφερθήκατε στον κύριο Κρόσεν. Ναι, ο κύριος Ρέινολτς μας είπε ότι ο κλάδος μπορεί να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τον καταναλωτή και συγκεκριμένα τους πιο νέου. Ναι, ευχαριστώ να απαντήσω, λέει ο κύριος Ρέινολτ. Ναι, αν θέλετε να ξεκινήσετε και κατόπιν θα παίρνει το λόγο η κυρία Φραντς και κατόπιν ε, η κυρία Στίκλερ και Βιλότα για την ε, προστασία, για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει ο κλάδος για να προστατεύσει κυρίως τους ανηλίκους. Ε, φυσικά είναι κριτική σημασία, ουσιαστική σημασία, ε, μία επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης και φυσικά διασφαλίζουμε με διάφορες διαδικασίες ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί και είναι κάπως δύσκολο όπως καταλαβαίνετε σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον γιατί δεν μπορούμε να τους δούμε. Υπάρχουν διαθέσιμες ορισμένες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη όπως ομάδα GB ε, και εκεί διατίθενται σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα των χρηστών και επαληθεύονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν επίσης για να χρησιμοποιήσει κάποιο πιστοτική κάρτα πρέπει να είναι άνω των 18. Υπάρχει λοιπόν μια ποικιλία ελέγχων που απαιτούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν μπαίνουν στην ιστοσελίδα μας επίσης. Ε, ε ε, συνασπισμός ε, φιλανθρωπίας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο απευθύνθηκε στον κλάδο για θέματα ασφάλειας του ηλεκτρονικού εμπορίου και είπαμε, υπόθηκε παραδείγματος χάρη ότι κάποια μέτρα που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο κλάδο θα πρέπει να αντιγραφούν και να εφαρμόζονται και σε περιπτώσει όπου έχουμε ηλεκτρονικό εμπόριο μόνο για ενηλίκους. Έτσι λοιπόν, ε, κανόνας προστασίας των δεδομένων ε, είναι πρόκληση για όλο τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όχι μόνο για τον κλάδο του τυχερών παιχνιδιών και επίσης το ψηφιακό θεματολόγιο. Μία από τις προκλήσεις είναι πώς μπορούμε να παληθεύσουμε την ταυτότητα των ανθρώπων πολύ γρήγορα. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό και δεν μπορούν να παίξουν τα παιχνίδια σου, τότε φυσικά θα πάνε αλλού. Και αυτή είναι μία από τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Προσπαθούμε να εξεύρουμε την ορθή ισορροπία. Δηλαδή πώ θα ταυτοποιήσουμε γρήγορα του ανθρώπου αυτού, πώ θα επαληθεύσουμε την ηλικία του και αφόσον μπουν στην ιστοσελίδα τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω. Αν ε, δεν έχουμε μπορέσει να επιβεβαιώσουμε 100% την ταυτότητα του ατόμου, δεν του επιτρέπουμε να αποσύρει χρήματα, ε, να αναλάβει χρήματα, αλλιώς ζητούμε φυσική ταυτότητα. Αν ε, στη συνέχεια ανακαλύψουμε ότι ήταν πράγματι ανήλικο το άτομο, τότε όλα αυτά τα χρήματα ε, θα επιστραφούν. Αν ε, το άτομο έχει χάσει αυτά τα χρήματα, τότε θα πρέπει να τα επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα, αλλά μάλλον κάποιο άλλο τα έχει κερδίσει. Έτσι λοιπόν αυτό μα κοστίζει χρήματα. Έχουμε κι εμεί λοιπόν χρηματοοικονομικό κίνητρο να διασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι δεν παίζουν τα δικά μα τυχερά παιχνίδια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φράντς. <laughs> Ähm, äh, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Σύντομα να εξηγήσω γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ πέρα από τη Σαξονία Άνχαλτ εκπροσωπώντας τα γερμανικά κρατήδια. Στη Γερμανία Έχουμε, όπως σας είπα, αυτή την σύμβαση μεταξύ των κρατηδίων για τυχερά παίγνια. Κάποια τυχερά παίγνια είναι αρμοδιότητα των κρατηδίων, αλλά συμφώνησαν σε αυτή τη σύμβαση τα κρατήδια και όπως σας είπα τώρα επεξεργάζονται μια νέα σύμβαση. Ε, ξέρετε πως ε, μας, μας αρέσει το ομοσπονδιακό μας σύστημα για το ερώτημα του κυρίου Κρόιτσμαν και βεβαίως ε, συστατικό τμήμα αυτού είναι η διάσκεψη των πρωθυπουργών των κρατηδίων που λαμβάνουν άρα αποφάσεις. Η Σαξονία έχει την τιμή φέτος να ασκεί την Προεδρία και να φιλοξενεί αυτή την διάσκεψη των Πρωθυπουργών, άρα εγώ είμαι επικεφαλής μιας ομάδας εργασίας που λέγεται το μέλλον του μονοπωλίου των τυχερών παιγνίων και άρα προετοιμάζουμε τις αποφάσεις των Πρωθυπουργών των κρατηδίων. Τώρα, πέρσι τον Οκτώβριο διάφοροι Πρωθυπουργοί είπαν πως αφενός θα πρέπει να διατηρηθεί το μονοπόλιο τυχερών παιγνίων, από την άλλη όμως να εξεταστούν διάφορα μοντέλα. Αυτά υποβλήθηκαν, αναπτύχθηκαν και το Μάρτιο του 2011 καταλήξαμε σε ένα άνοιγμα με άδειες στο στοίχημα το αθλητικό. Κατόπιν υπήρχε μια άλλη ειδική διάσκεψη στην οποία ε, την οποία ανέφερε ο κύριος Κρόιτσμαν και εκεί πέρα, εκεί το κρατήδιο του Σλέσφι Χόλσταν δεν συμφώνησε με την υποβληθήσα πρόταση και η κατάσταση τώρα έχει ως εξή. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα επιτάπητος. Εγώ είμαι πεπισμένη πως είναι ισχυρός ο φεντεραλισμός στη Γερμανία και θα βρεθεί μια κοινή λύση. Τα δε κρατήδια θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται αυτή την πρότασή τους και προετοίμασαν στις 6 ε, Τετάρτου όπως σας είπα αυτή την πρόταση και ε, επ' αυτού εργαζόμαστε. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ενδιαφέρει όλη αυτή η εσωτερική κατάσταση. Α, τέλος, ε, για το ερώτημα αυτό, το τι θα γίνει με το Schleswig Holstein, κοιτάξτε, εμείς συνολικά, όπως σας είπα, θα συνεχίσουμε με την πρότασή μας αυτή και νομίζω πως μεταξύ των ε, κρατηδίων θα λάβουν χώρα συζητήσεις και ε, γνωρίζουμε όλοι την ευθύνη που φέρουμε. Η παρατήρηση τώρα πως ε, η απόλυτη απαγόρευση στο ίντερνετ δεν οδηγεί πουθενά οδήγησε αυτό και από την δική μας σκοπιά στο να αναγνωρίσουμε πως ε, υπάρχει μια σοβαρή παράνομη αγορά και με τις διατάξεις στη νέα μας πρόταση προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε αυτό με ένα προσεκτικό άνοιγμα της ε, αγοράς δηλαδή το λέμε απαγόρευση με μια επιφύλαξη δότησης όπως σας είπα, για, αυτό το, για κάποια είδη στοιχημάτων. Οπότε απομακρυνόμαστε κάπως από την απόλυτη απαγόρευση. Τώρα για το θέμα που ανέφερε πάλι ο κύριος Κρότσμαν για το πώς θα γίνει η επιλογή 7 ε, εταιριών μόνο να λάβουν άδειες. Εμείς προβλέπουμε ένα σύστημα στο οποίο δεν θα υπάρχει ε, ένας απεριόριστος αριθμός αδειών, αλλά θα είναι περιορισμένος και αυτό γιατί δεν σκοπεύουμε η αγορά μας να επεκταθεί. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μαύρης αγοράς και να το διοχετεύσουμε κάπως. Και είμαστε πεπισμένοι πως ε, η ρύθμιση αυτή που προβλέπουμε που μπορεί να τη μελετήσει ο καθένα, θα οδηγήσει στο να βρούμε τους κατάλληλους, τις κατάλληλες εταιρείες. Ε, θαυμάζουμε την αισιοδοξία σας εδώ στο Προεδρείο, κύριο Στίκλε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Πρώτον, θέλω να αυτοσυστηθώ όχι ως εκπρόσωπος μονοπωλίων, γιατί έχουμε και μέλη με απελευθερωμένες αγορές. Από την Ιταλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μέλη. Καλύπτουμε ολόκληρο το φάσμα. Τώρα, το πιο κρίσιμο θέμα. Όταν ε, συζητούμε για ε, παράνομη ή μη εγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών από επανέρχομαι σε αυτά που είπα στην αρχή μου παρουσίαση. Το πλέον σημαντικό ζήτημα είναι η εφαρμογή του νόμου. Μπορείτε να έχετε έναν αδιούχο, 7 όπως ε, προετοιμάζει η Γερμανία ή εκατοντάδες όπως η Ιταλία. Το θέμα είναι να προστατεύονται οι φορολογούμενοι και να εφαρμόσετε σωστά ο νόμος. Ε, γιατί ε, η χαμηλή φορολογία είναι το πρόβλημα αυτής της αγοράς αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε για λαχιοφόρους αγορές και εδώ επισέρχεται και το κοινωνικό μοντέλο που συζητούσαμε, δεν είναι υψηλό το ποσοστό όταν, ε, ε, ε, φορολογι... όταν δίνεται ως φόρος κάτω από το 1% του τζίρου καταλαβαίνετε ότι προσελκύονται εύκολα οι παίκτες και παρασύρονται. Ε, ε, δηλαδή μπορεί να έχετε νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης αδειοδοτημένους, μπορείτε να έχετε κάποιους φορείς που έρχονται από την Καραϊβική ή από τη Λατινική Αμερική, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή επιβολή του νόμου. Αν δεν υπάρχει αυτό, ούτως ή άλλως ε, θα προσανατολίζονται όλοι προς παράνομες αγορές γιατί υπάρχει υψηλότερη κερδοφορία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για καλούς σκοπούς. Μπορείτε ε, να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα, τους φόρους ή αλλιώς θα έχετε μία ανοιχτή αγορά ε, με ε, κέρδη 90-95%. Το θέμα είναι η προστασία των παικτών και όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε. Θα ήθελα να καλύψω εν συντομία μια άλλη ερώτηση. Το betting right, το δικαίωμα του στοιχηματίζειν είναι ένα και ο συνδυασμό του με ε, τα πνευματικά δικαιώματα. Πέραν της Γαλλία δεν υφίσταται νομική βάση για ε, καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά η αγορά των ε, λαχείων αναγνωρίζουν φυσικά την ανάγκη συμβολής από πλευρά του παρόχου των στοιχημάτων στην χρηματοδότηση της λαχιοφόρου αγοράς, αλλά δεν θέλουμε να επιβληθεί ένα φόρο για τους διοργανωτές των αθλητικών συναντήσεων γιατί έτσι θα συγκεντρωθούν χρήματα μόνο σε λίγα αθλήματα, ε, ελάχιστου συνδέσμου. Έχουμε πάνω από 200 ε, στην Ευρώπη. Δεν νομίζω να ε, τελεσφορήσει η λύση. Εγώ φαντάζομαι ένα διαφορετικό πρότυπο, δηλαδή συμβολή για να την αλληλεγγύη, για τη διαφάνεια. Τα χρήματα που συλλέγονται μπορούν να αναδιανέμονται από μη κερδοσκοπικέ αθλητικέ ενώσει. Παραδείγματο χάρη στην Αυστρία έχουμε ένα αντίστοιχο Έχουμε την, ε, μια τέτοια οργάνωση που κατανέμει τα χρήματα. Φυσικά το ποδόσφαιρο παίρνει τα περισσότερα κονδύλια γιατί έχει και τα περισσότερα στοιχήματα, αλλά όχι μόνο. Ε, για λόγους αλληλεγγύης κατανέμουμε τα κονδύλια και σε άλλα αθλήματα. Αυτά λοιπόν, ε, ε αυτή, είναι το σημαντικό από πλευρά του νομοθέτη για το θέμα του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Ε, διακρίνω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν ε, μιλάμε ε, για το ξέπημα βρώμικου χρήματος, εγκληματικότητα και στήσιμο αγώνων. Θα σας υποβάλουμε σχόλια για την πράσινη βίβλο και θα τα αναφέρουμε αυτά εδώ. Οπωσδήποτε πρέπει να αναλυφθεί η δράση. Ο μπορεί να χάσει την κεραιότητά του ο χώρος του αθλητισμού. και ε, θα έχουμε τρομακτικές εξελίξεις. Ε, οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να αποδοθεί ιδέουσα σημασία σε αυτό το στοιχείο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρέινολτς θέλει να επανέλθει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε τον κύριο Βιλότε πρώτα και μετά αν έχετε κάτι σύντομο, κύριε Ρέ. Ευχαριστώ να επανέλθω στο θέμα της ε, ακεραιότητας του ήθους και το δικαίωμα του στοιχηματίζει. Είναι εντελώς ε, διαφορετικό θέμα της επιστροφής του τομέα στο σύνολό της. Ε, γι' αυτό υπάρχουν μηχανισμοί, παραδείγματος χάρη φόρου, όταν έχουμε στοιχήματα. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται αυτό που θίξατε. Τώρα το δικαίωμα του στοιχηματίζει είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Είναι μια νομική έννοια που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά τη διάδοση τη εικόνα. Ε, Κανένα ε, φορέα διάδοση ε, δεν θα ε, διέδιδε μια εικόνα χωρί να έχει έρθει σε πρώτερη συμφωνία με το διοργανωτή. Γιατί μιλάμε για το δικαίωμα τη άειλη ιδιοκτησία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα στοιχήματα. Αν κάποιο οργανωτή θέλει να προτείνει στοιχήματα για ένα αθλητικό γεγονό, θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία εκ των προτέρων με τον οργανωτή του αθλητικού γεγονότου τη αθλητική εκδήλωση. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε ε, και ε, αυτό το φελός Έχουμε και το όφελος του οργανωτή αλλά και ένα ηθικό σκέλος γιατί μπορεί ο διοργανωτής να έχει πρόσβαση στο ποσό των στοιχημάτων που έχουν καταγραφεί από την ε, ιστοσελίδα των στοιχημάτων γιατί διαφορετικά ε, ε, είναι στα τυφλά. Δεν μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο της αθλητικής εκδήλωσης που οργανώνει. Χρειάζεται λοιπόν ένας πλήρης μηχανισμός, χρειάζονται υποχρεωτικές νομικές σχέσεις μεταξύ του που Επίση, στο σελίδα και του διοργανωτή, μαζί ε, με ε, τη συμμετοχή των αρμοδίων δημοσίων αρχών και φυσικά εκεί μπορούν να παρέμβουν οι δημόσιες αρχές. Χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζονται και αθλητικές κυρώσεις αλλά και ποινικέ κυρώσεις. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο ε, για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν μιλάμε για κάτι διαφορετικό θετικό εδώ από τη χρηματοδότηση ε, του αθλητικού κλάδου. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα δύο αυτά ζητήματα. Τώρα, σε σχέση με την ηχληλασιμότητα ε, του σεβασμού της ηλικία και της καταπολέμησης της νομιουποίησης παράνομων εσόδων. Το σύστημα που έχει συσταθεί στη Γαλλία, ε, όταν ανοίγει ένας παίκτη ένα λογαριασμό, υποχρεώνεται να υποβάλει αντίγραφο της ταυτότητάς του και αυτό το αντίγραφο το διατηρεί στην κατοχή της η ρυθμιστική αρχή. Έτσι λοιπόν ο παίκτη, εφόσον ε, έχει δώσει μαρτυρία της ηλικία τους και θα πρέπει να δώσει ε, τα στοιχεία ενός λογαριασμού πληρωμής που θα έχει ε, ανοίξει από τον ίδιο, θα έχει ανοιχθεί από τον ίδιο το χρήστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν η ρυθμιστική αρχή μπορεί να ελέγξει ανοίξει αυτό το συγκεκριμένο λογαριασμό. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει διαφάνεια ακριβώς για να καταπολεμήσουμε την ομοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες εγκληματικέ δραστηριότητες. Sorry. Ε, Ίσως θα μπορούσε ε, ο κύριος Ράινερς να απαντήσει και στο δικό μου ερώτημα. Uh, ναι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρέινολτς ε, πολύ σύντομα. Ναι, αν μου επιτρέπετε αν ε, απαγορευτεί, ε, αν απαγορευτεί τα τυχερά παιχνίδια δεν υπάρχει διανομή και είπατε στην περίπτωση που δεν υπάρχει ρύθμιση στις χώρες τι γίνεται με τα κέρδη. Δηλαδή για τη φορολόγηση των κερδών, με ρωτήσατε. Αυτή είναι μια απόφαση που θα αντιλάβουν οι κυβερνήσει. Αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να φορολογείται το κέρδο ενό ατόμου, τότε εντάξει και φυσικά ε, οι εταιρείε θα πρέπει να το σεβαστούν αυτό. Σε ορισμένα μέρη ε, του πλανήτη υπάρχει τέτοια φορολόγηση των κερδών, ενώ σε άλλα μέρη όχι. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατανομή για ε, κοινό όφελο, ε, παραδείγματο χάρη, ακούσαμε εδώ ότι πρέπει να υπάρχει μια αναλογία. Το μοντέλο τη λαχιοφορού αγορά είναι ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο. Ε, το, η αναλογία τη εξόφληση τη πληρωμή είναι εντελώ διαφορετική. Για, έτσι λοιπόν, η δυνατότητα τη λαχιοφορού να συνεισφέρει σε πληρωμή για καλό σκοπό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι λοιπόν εμείς, ε, αν μας βάλετε ε, σε αυτή τη διαδικασία, είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο καταναλωτή. Δηλαδή, αν αναγκάσουμε τον καταναλωτή να πληρώσει υπερβολικά για ένα προϊόν που μπορεί να το βρει αλλού, ξέρετε τι θα γίνει, θα πάει αλλού ο καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά όσα είπε η κυρία Κορόλα, γιατί το χάρη δεν προστατεύουμε το χάρη το, και δεν κάνουμε κάτι ε, με το θέμα των πολλαπλών ε, λογαριασμών. Ξέρετε, ε, ε εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί ένα άτομο να έχει πολλά απλούς λογαριασμούς γιατί παίρνουμε ένα αποτύπωμα του υπολογιστή του ατόμου. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς λογαριασμούς και να μπει από πολλαπλούς λογαριασμούς στην ιστοσελίδα. Ε, έχουμε επίσης πάρα πολλές μελέτες και από τον καθηγητή Μάικλ Λίβι από το Πανεπιστημίο του Κάρντιφ, ε, ο οποίος είναι και συνεργάτης της ε, Βρετανικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό και διερεύνησε το θέμα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μας των τυχερών παιχνιδιών και ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει εκτεταμένος τέτοιο κίνδυνο. Πρόεδρος. Ναι, ε, ακούσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικέ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τμήμα. Έχουμε τον κύριο Μάικλ Μπέι Γιόρσελ, ελπίζω σωστά να πρόφερα το όνομά σας, είναι ε, επικεφαλής ε, του κέντρου ε, για τον ε, εθισμό στο τυχερά παιχνίδια της Δανίας. Έχουμε τον κύριο Τρέβορ Ντέιβιτ από το Gum Care, θα μας εξηγήσει τι συνιστάτη αυτή η οργάνωση του Ηνωμένου Βασιλείου, που επικεντρώνεται στο προβληματισμό, στο, συγγνώμη, στο... Ε, παθολογικό τζόγο. Επίση έχουμε τον κύριο Πέρα από την Φιλανδία, από την οργάνωση ΡΕΙ, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, αξιωματούχος του RAY. Ε, θα μας ενδιαφέρει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι κάνουν σε σχέση με την τεχνολογία. Και τέλος, τον κύριο Ματιέ Μορέη, ο οποίος εκπροσωπεί την Βρετανική Λίγκα θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιόρσελ, ο οποίος ε, έχει πέντε λεπτά στη διάθεσή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε τις διαφάνειες. Θα ήθελα να κάνω μία σύντομη παρουσίαση του κέντρου ε, παθολογικού τζόγου Στη συνέχεια θα κάνω σχόλια για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση και μετά θα με μιλήσουμε για την προστασία των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα κέντρο για τους εθισμένους στο τζόγο. Ιδρύθηκε το κέντρο το 92 και είμαστε το παλαιότερο και μεγαλύτερο τέτοιο κέντρο για τον παθολογικό τζόγο, τους παίκτες και τους συγγενείς τους. Ε, ε, λειτουργούμε σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Ε, περίπου φέτος, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, είχαμε 1.500 πελάτες, παίκτες, οικογένειες εκεί και ομάδες υποστήριξης. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Οι βασικοί τομεί δραστηριότητα είναι η θεραπεία, η πρόληψη και η έρευνα. Ε, εδώ και εξώνοσοκομιακή θεραπεία, παρακολούθηση, ομάδε υποστη... ψυχολογική υποστήριξη κτλ. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Το 2008 ε, κάναμε Φτιάξαμε μία εκτεταμένη ιστοσελίδα προσβάσιμη και στους μαθητές και στους ανηλίκους και χρησιμοποιείται ευρέω στα σχολεία και έχουμε διεξαγάγει μελέτη κατά όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κέντρου. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, έχουμε ε, τα στοιχεία για το 2008 οι νέοι πελάτες είναι 314 και 2,2% από τους 314 νέοι πελάτες απάντησαν καταφατικά στο ερώτημα αν ε, παίζουν τυχερά παιχνίδια και κυρίως σε απευθεία σύνδεση. Για πέρσι έχουμε τον αριθμό των νέων πελατών που εκτινάσεται στο 936 και το 44% παίζουν μόνο σε απευθεία σύνδεση. Ε, πρόκειται για ε, ε, τεράστια άνοδο, αλλά αυτό δεν ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια της Δανίας βάσει των στοιχείων του κέντρου. Τι, ποια είναι αυτά τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση. Το πόκερ είναι πρώτο στη σειρά με ποσοστό 44% μετά τα στοιχήματα και μετά τα φρουτάκια. Επόμενη διαφάνεια ο πραγματικός κόσμος και ο εικονικός κόσμος. Έτσι το διαδίκτυο, αυτό είναι το θέμα μας, σχεδόν εξισώνονται ως προς τη διανομή και σε λίγα χρόνια το διαδίκτυο θα καταλάβει την πρώτη θέση ε, ε, στα τυχερά παιχνίδια και ε, ο πραγματικός κόσμος θα πέσει το 30-35% κατά τη γνώμη μου, γιατί έχει τόσο πολλές δυνατότητες να προσφέρει το διαδίκτυο που δεν προσφέρονται από, τις παραδοσια... από τα παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια. Προσφέρεται επίσης απόλυτη διαθεσιμότητα. Για λίγο μπορείτε να παίξετε ανώνυμα, είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση σε περισσότερα χρήματα αν αργά το βράδυ είσαστε μπροστά μπροστά στον υπολογιστή σας ε, και δελεάζεστε γιατί ξέρετε ότι μπορείτε εύκολα να δανειστείτε χρήματα από κάποια τράπεζα και να παίξετε. Υπάρχουν κάποιοι ε, που παίζουν ολόκληρη τη νύχτα, 24 ώρες το 24 μπορείτε να παίζετε αν θέλετε. Επόμενη διαφάνεια ε, για τα, την απευθείας σύνδεση το ε, χρησιμοποιούνται οι διαδικτυακοί τόποι σε ποσοστό 90% από πλευρά ε, των δανών. Τώρα για τα στοιχήματα. Είναι υπέρ των καταναλωτών. Δεν ξέρει κανεί με σιγουριά. Έχουμε μεγάλο ποσοστό παθολογικού τζόγου και κυρίω εναγνία των ίδιων των παικτών σε πολλέ ε, περιπτώσει κάτω από 100.000 ε, δανεί με ε, διαφορετικούς τρόπους είχαν προβλήματα με τον τζόγο ε, το 2010 και ελπίζω να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το 2012 και να έχουμε παρκή στατιστικά στοιχεία ώστε να κάνουμε και συγκρίσει. Ένας παλιό ήρωάς μου είναι ο Μπομπ Ντίλαν και τραγουδούσε ε, λέγοντας ότι υπάρχουν αλλαγές, οι καιροί αλλάζουν και ελπίζω το ίδιο να γίνει και για τα τυχερά παιχνίδια. Η νέα νομοθεσία στη Δανία ευελπιστούμε ότι θα εμφανιστεί τον Ιανουάριο του 2012. Εν μέρει απελευθερώνεται η αγορά των παιχνιδιών στη Δανία και καλωσορίζουμε κατά τη γνώμη μου την πραγματικότητα. Η νέα νομοθεσία ε, προτείνει λογικά μέτρα για να ελεγχθεί η αγορά των τυχερών παιχνιδιών και να δεχτούμε το τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο προσφέροντας ε, υπηρεσίες για συγκεκριμένες ε, πληθυσμιακές ομάδες γιατί αυτό χρειαζόμαστε στη Δανία. Ευχαριστώ. Thank you very much for that Εμείς σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε όλες αυτές τις γνώσεις μαζί μας ε, και ο κύριος Ντέιβιτ τώρα. Hello Γεια σας. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Λέγομαι Τρέβορ Ντέιβιτ. Εργάζομαι για την Care μια εθνική κοινοφελή οργάνωση. Παίζουμε διπλό ρόλο, δηλαδή συνεργαζόμαστε και με τον κλάδο του τζόγου και τους εκπαιδεύουμε σε εταιρική κοινωνική ευθύνη κτλ. Έχω δύο μόνο διαφάνειες για να σας δώσω μια γεύση των ε, εμπειριών μου δίνω και συμβουλές και εκπαιδεύω άλλους συμβούλους. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι πως ε, ο τζόγος είναι ένα προβληματικό, ένα πολύπλοκο με ζήτημα. Ο δε τζόγος στο ίντερνετ έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κινδύνους και αυτό το οποίο βλέπουμε με τους προβληματικούς παίκτες είναι πως ε, τζογάρουν σε πολλές δραστηριότητες δεν χρησιμοποιούν μόνο το διαδίκτυο, πάνε και σε μαγαζιά και σχηματίζουν και σε άλλες δραστηριότητες. Οπότε το πρόβλημα είναι ο τζόγος και όχι η δραστηριότητα στην οποία λαμβάνουν μέρος. Βεβαίω υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, η ταχύτητα του στοιχήματο και η ταχύτητα τη πληρωμής, που τα ξέρουμε. Μετά. Έχουμε δει μια κάποια βελτίωση γιατί έχουμε και εμείς νούμερα ε, με το πρόβλημα και το διαδικτυακό τζόγο και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο φίλων. Έχουμε δει μια αύξηση νομίζω της 100 ε, των γυναικών στο διαδικτύο, το οποίο έφτασε 23% πέρσι, οπότε ε, βλέπουμε πως οι ευπαθείς ομάδες είναι οι γυναίκες και οι νέοι που φαίνεται να προτιμούν ε, το τζόγο στο διαδίκτυο και η προσέγγιση που έχουμε είναι πως χρησιμοποιούμε ένα κοινωνικό μοντέλο κοινωνικού αντικτύπου εργαζόμαστε με τους ανθρώπους που επηρεάζονται από ένα προβληματικό παίκτη οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 15 άτομα οικογένεια, φίλοι, παιδιά, εργοδότες κτλ. Οπότε έχουμε ένα τέτοιο μοντέλο και αντιμετωπίζουμε το, τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και τι κάνουμε. Έχουμε μια προσέγγιση κοινωνικής ευθύνης, δηλαδή πηγαίνουμε σε οργανώσεις όπου μπορεί να συναντήσουμε προβληματικούς παίκτες, τους εκπαιδεύουμε, τους ενημερώνουμε για τα σημάδια του προβληματικού τζόγου και Εργαζόμαστε βεβαίω ε, και συνεργαζόμαστε και με άλλους επαγγελματίες, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Επόμενη διαφάνεια. Το άλλο μισό των δραστηριοτήτων μας είναι η συνεργασία με τον κλάδο και αφορά την κοινωνική ευθύνη όσα έχετε συζητήσει δηλαδή ε, στην Πράσινη Βίβλο συζητάμε ταυτοποίηση της ηλικία και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο εκπαιδεύουμε ε, ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα αυτών, αυτών και online επίσης και κάνουμε και διεθνείς διαβουλεύσεις. Να συνοψίσω το τι κάνουμε λοιπόν. Συμφωνώ με την αποστολή της οργάνωσής μας. Εμείς δεν κρίνουμε αυτό το οποίο κάνουμε είναι το, τι γίνεται όταν κάποιο έχει πρόβλημα με τον τζόγο και θέλουμε ακριβώ αυτή την αντίληψη να βελτιώσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ανοίξει ο τζόγο, ε, ειδικά στο διαδίκτυο, πρέπει να εκπαιδευτούν όχι μόνο οι χρήστε, οι ίδιοι οι παίκτε, γιατί το στατιστικό αυτό στοιχείο του 75, 85% του τζόγου που είναι χωρίς άδεια στο διαδίκτυο είναι ακριβώς, ε, δείχνει τη σημασία του το ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους καταναλωτές. Και όταν ε, ενημερώνουμε εμεί κάποιον θα κάνει ένα site κάτι. Ε. Επίσης το ίδιο και για ξένες αρχές. Το να εκπαιδεύουμε λοιπόν τους καταναλωτές να αναζητούν αυτό το σηματάκι, να ξέρουν ότι σχηματίζουν με ασφάλεια. Και να προωθήσουμε μια υπεύθυνη προσέγγιση στο, απέναντι στο τζόγο, ερευνούμε περαιτέρω και υποστηρίζουμε, όπως σας είπα, πρωτοβουλίες εταιρική ε, κοινωνικής ευθύνης ε, στον τομέα του, των τυχερών παιχνιδιών. Αυτά κάνουμε. Ευχαριστώ που μιλήσατε ακριβώς 5 λεπτά, ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο κύριος τώρα Περάκυλα που θα μας πει για τις εμπειρίες σας με την προστασία παικτών και το διαδικτυακό παιχνίδι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξαιρετικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπω κατευθείαν. Η φιλανδική κυβέρνηση μας ε, έδωσε μας ε, ανέθεσε να δημιουργήσουμε ένα καζινό για τους φιλανδούς πλέκτες, μια υπηρεσία τυχερών παιχνιδιών για τους φιλανδούς πλέκτες. Ε, η δουλειά γίνεται εκεί και θα σας ε, παρουσιάσω τα κύρια στοιχεία της εργασίας μας και ελπίζω να προβληματιστείτε έτσι ώστε να προωθήσετε τα πράγματα τώρα, ταυτοποίηση των παικτών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλουμε να μιλήσουμε για μεγάλες προκλήσεις ε, από τη Σκοπιά ε, της ε, ταυτοποίησης ε, των πελατών και της νομοποίησης παράνομων εισόδων. Εδώ. Βλέπετε πως υπάρχει διασκορπισμός των δραστηριοτήτων σε διάφορες χώρες αυτό το θέμα σχετίζεται και με την ε, Πράσινη Βίβλο και με την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων Δηλαδή, τίθεται το θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα και πώς θα διασφαλίσουμε ότι σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια των διασυνοριακών δραστηριοτήτων ε, μπορούμε να προβαίνουμε σε ταυτοποίηση των πελατών και πώς ε, μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις. Πώς μπορούμε ε, να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του παίκτη, του πελάτη ε, κάποιος ε, μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας ε, μόνο κάποιους κωδικούς ταυτοποίησης ηλεκτρονική, ηλεκτρονικού banking έτσι λοιπόν, όταν ανοίγει κάποιο ένα λογαριασμό, αμέσω ε, σε πραγματικό χρόνο γίνεται ταυτοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία τη Φιλανδία. Εγώ μπορώ να σα πω ότι επίση παίζω τυχερά παιχνίδια και το να δημιουργήσει κάποιο ένα λογαριασμό στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί παραδείγματο χάρη να αγοράσει ένα eBay box ε, που κοστίζει πάρα πολύ φθηνά και μπορεί να αλλάζει ο παίκτη, παραδείγματο χάρη κάθε 15 λεπτά, την διεύθυνση του eBay για να κρύβει την ταυτότητά του. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ταυτοποιούμε τον πελάτη. Επίση μπορούμε να ε, βλέπουμε ποια είναι η ηλικία του ατόμου μέσω του Εθνικού Μητρώου και ε, ποια είναι και η οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή ποιος έχει την κυδαιμονία. Είναι αδύνατο στη Φιλανδία ε, να παίξει τυχερά παιχνίδια κάποιος ανήλικος. Έτσι λοιπόν προστατεύουμε τις ευάλωτες ομάδες. Βέβαια, όταν μιλάμε για ευάλωτε ομάδε, δεν μιλούμε μόνο για του ανηλίκου, αλλά μιλάμε και για ανθρώπου οι οποίοι ε, δεν είναι σε θέση να παίξουν. Παραδείγματο χάρη, ε, εμείς χρησιμοποιούμε ένα σύστημα που βλέπουμε ε, αν ε, το άτομο αυτό, παραδείγματο χάρη, έχει μια πιστοτική κατάσταση που του επιτρέπει να παίξει ή όχι. Έτσι λοιπόν ε, προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει να καταβολμήσουμε αυτές τις καταχρήσεις ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχουμε μπόνους ε, για τις καταθέσεις, ούτε δίνουμε μπόνους στους παίκτες σε σχέση με τον όγκο των κερδών τους. Έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο εργαζόμαστε κατά των δικών μας συμφερόντων γιατί αυτή είναι η παραδοσιακή τρόπη να παγιδεύσει κάποιους τους παίκτες. Όμως εμείς δεν εφαρμόζουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε νομοθεσία στη Φιλανδία, η οποία αποτελεί τη βάση και επίσης έχουμε και ένα εργαλείο play scans, άρρωσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τον παίκτη για τη δική του συμπεριφορά. Έτσι, λοιπόν, στη Φιλανδία τους τελευταίους 6 μήνες παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίε και θεωρούμε ότι δεν χρειαζόμαστε συστάσεις, αλλά χρειαζόμαστε πραγματική ρύθμιση, πραγματική νομοθεσία και πραγματική εποπτεία και έλεγχο. Δεν χρειαζόμαστε πλέον συστάσεις. Και η ιδέα ότι ένα άτομο μπορεί να έχει μόνο ένα λογαριασμό για να παίζει είναι κάτι που θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα πραγματικά δεδομένα του όγκου ε, του τζόγου και έχουμε και τα πραγματικά στοιχεία για τους παίκτες. Και ο Σκορμπή είπε πόσο πολύ δύσκολο είναι να έχουμε στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα. Έτσι λοιπόν ε, βλέπετε ότι λείπουν οι πληροφορίες και έχουμε και αυτό το πρόβλημα στη Φιλανδία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι και πάλι επανερχόμαστε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τελευταίος ομιλητής ο κύριος Μορέγη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά, διότι εκπροσωπώ σήμερα ε, την οργάνωση κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, έχουμε 40 περίπου μέλη αθλητικών ενώσεων από διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και διεθνών ενώσεων για διάφορα αθλήματα. Ελπίζω, ελπίζω να τα καταφέρω μέσα στα λίγα λεπτά που δικαιούμαι. Ούτω ή άλλω έχουν υποθεί τα περισσότερα από αυτά που θέλαμε να πούμε, οπότε απλοποιείται το έργο μα. Τρει παρατηρήσει ε, θα κάνω για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το ήθο, η ακαιρεότητα του αθλήματο. Ε, αυτό αφορά τι αθλητικέ ενώσει, φορεί εκμετάλλευση και του καταναλωτέ. Τρει παρατηρήσει θα κάνω και θα κάνω και δύο προτάσει, δύο συγκεκριμένα μέτρα στα πλαίσια τη εκθέση του κυρίου Κρόιτσμαν. Τρει παρατηρήσει πρώτα απ' όλα τα στοιχήματα δεν δημιούργησαν το στήσιμο αγώνων ε, και τις απάτες. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό νομίζω. Τα στοιχήματα ε, δεν είναι η πηγή ε, ούτε και η απόρρια όλων των δεινών του αθλητισμού όπως τα γνωρίζουμε σήμερα και όπως ήταν ανέκαθεν ούτως ή άλλως. Ε, με την, ε, το διαδίκτυο υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στοιχημάτων και απλώς πολλαπλασιάστηκαν οι κίνδυνοι που συνδέονται ε, με τα στοιχήματα. Στην αρχή στοιχηματίζαμε, ας πάρουμε το ποδόσφαιρο για την ομάδα που θα κέρδιζε τον αγώνα ή για τον αιτημένο. Σήμερα μπορούμε να στοιχηματίσουμε για τα πάντα. Ε, Πώ θα γιορτάσει ένας ποδοσφαιριστής ε, όταν βάλει γκολ, αν θα στριφογυρίσει τρει φορέ ή θα βγάλει τη φανέλα του ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλέ εκδηλώσει, πάρα πολλά συμβάντα ε, που μπορούν να οδηγήσουν σε στοιχήματα. Όλα τα αθλήματα δεν καλύπτονται, κανένα δεν είναι προφυλαγμένο και οι μελέτε δείχνουν ότι τα λιγότερα εκτεθειμένα αθλήματα είναι τα μικρή κλίμακα. ας τα πούμε έτσι, τα ίσονο σημασία αθλήματα. Ε, αλλά δυστυχώ διατρέχουν αυξημένου κινδύνου. Στο Μάντσεστερ το Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ έχει κάνει μια ε, κατατοπιστικότατη μελέτη για αυτό το θέμα, αλλά επιμένω ε, για του αυξημένου κινδύνους για τα μικρά αθλήματα. Δεύτερον, το ήθο στον χώρο του αθλητισμού έχει κέρια σημασία, όπω είπα, για όλου του φορεί, για του φορεί για τι λαγιοφόρου αγορέ για τι αθλητικέ ενώσει και προφανώ για του καταναλωτέ, διότι όταν στείνονται οι ε, οι καταναλωτέ χάνουν χρήματα, το ίδιο και οι φορεί. οι καταναλωτέ καταναλωτέ ε, ε, ενδέχεται να χάσουν και την εμπιστοσύνη τους ε, στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και οι διοργανωτές ω εκ τούτου δεν θα πολλούν με εξίσου καλά, αν θέλετε, τις συναντήσεις τους. Και υπάρχει και ένα εμπορικό συμφέρον, γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς, πρέπει να διαφυλάξουμε το ήθος του αθλητισμού. Ε, τι κάνουμε λοιπόν για να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι αθλητικές ενώσεις ε, θέσπισαν συστήματα επιτήρησης ε, ή διορισμού τελευταία στιγμή του διαιτητή κάθε αγώνα, απαγόρευση στοιχημάτων ε, για, τα για κάποια μέλη των αθλητικών ενώσεων. Μία πληθώρα μέτρων που έχουν θεσπιστεί είναι σχετικά αποτελεσματικά αλλά και επισύρουν μεγάλο κόστος ταυτόχρονα στη δική μας ένωση δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά για αθλήματα λιγότερο, που δεν είναι τόσο πολύ στο φως της δημοσιότητας, αν θέλετε, λιγότερο ε, ακριβά ε, σε εισαγωγικά αθλήματα, το κόστος επιβολής των μέτρων ε, είναι απαγορευτικό. Οπότε είναι σημαντικό το οικονομικό διακύβευμα για κάποια αθλήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μας, πρώτον, ε, μέσα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θέλαμε να συμπεριλάβετε το εξή, ε, την, αναγνώριση, την έννοια τη αναγνώριση ε, τη απάτη σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τουλάχιστον μία σύσταση για την αναγνώριση τη απάτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί, διότι θα μπορούσαμε να συντονίσουμε τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων, των ενδίκων μέσων που διαθέτουμε για να καταπολεμήσουμε τι συχνά διασυνοριακέ παραβάσει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προβλέπεται ήδη το ίντρανετ το έχουμε στη Γαλλία. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλαμε να ασκήσει πίεση, ούτως ώστε όχι να καταλήξουμε σε εναρμόνιση απαραίτητα, αλλά τουλάχιστον ε, να έχουμε ένα είδος συντονισμού για τον ορισμό ε, της ε, αθλητικής απάτης. Και δεύτερον, που συζητήθη, ένα θέμα που συζητήθηκε εκτεταμένα, το δικαίωμα το στοιχηματίζει ή αυτό που εγώ ονομάζω νομικά δεσμευτικές συμβατικές σχέσεις. Ο κύριος Βιλότα αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσαν πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι σημαντικό αυτό κυρίως για το ποδόσφαιρο. Όχι ότι είναι πνευματικό το ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο, έτσι, αλλά μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα. Είναι εντελώ διαφορετική έννοια. Το δικαίωμα λοιπόν ε, για να ε, βάζει κάποιο στοιχήματα ή το θέμα των ε, συμβάσεων που θα είναι νομικά δεσμευτικέ έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι έτσι οι αθλητικέ ενώσει υπό την εποπτεία των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων εκμεταλλεύσεων μπορούν να προσδιορίσουν τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε του τιμένου αγώνε. Επίση προσδιορισμό των εγκεκριμένων και μη στοιχημάτων και επ' αυτού νομίζω ότι είναι βασικό ο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι αθλητικέ ενώσει διότι για ορισμένα στοιχήματα είναι ανέφικτο να οργανωθεί νομίμως ε, το σύστημα στοιχημάτων. Ο μαραθώνας ε, του Λονδίνου, ε, ο μαραθώνιος <laughs> συγγνώμη, του Λονδίνου έχει απαγορεύσει τα στοιχήματα παραδείγματο χάρη. Πρέπει να ακουστεί η φωνή των αθλητικών ενώσεων και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να ασκήσει την πίεση που σας δίσαμε προηγουμένως. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. πολύ καλές οι συστάσεις, οι προτάσεις σας και ευχαριστούμε για την ανασκόπηση. Έχουμε ε, χρόνο. Θέλω να ακούσουμε και την κυρία Πρόεδρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακούσουμε και τη σύνοψη του εισηγητή. Α ακούσουμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη και την κυρία Σάλτεμόζη. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το παίρνω σαν δεδομένο ότι όλοι συμφωνούμε πω τα τυχερά παιχνίδια, ο τζόγο, είτε διαδικτυακά είτε όχι, ενέχουν τον κίνδυνο εθισμού και πολλές φορές οδηγούν και σε παρεμφερή προβλήματα. Η εμπούλωση του προβλήματος επιτυχάνεται όταν πρώτα αναγνωρίσουμε το ίδιο το πρόβλημα. Συνεπώς το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τη λειτουργία των επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών είτε επιτρέπει την ύπαρξη και δραστηριοποίηση ιδιωτικών εταιριών είτε όχι θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όσοι απαρτίζουν την αγορά ακολουθούν πολύ υψηλά πρότυπα κοινωνικής ευθύνης. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρακτικές εντοπισμού και διαχείρισης των εθισμένων παιχτών, αναλύοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συχνότητα επισκέψεων, τον τρόπο παιχνιδιού, τη στρατηγική για κέρδη, μπορούν να εντοπίζονται οι εθισμένοι χρήστες και να τους διοχετεύεται πληροφορήση για συμβουλευτική αγωγή. Η ερώτηση μου επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτή την υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης κατά πόσο τέτοιες ρήτρε μπορούν να τεθούν ως προαπαιτούμενο για την ύπαρξη και λειτουργία των εταιριών στο διαδίκτυο. Είναι έτοιμη η επιχειρηματική κοινότητα να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές ως βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Uh, Ευχαριστώ, η κυρία Ευχαριστώ. Θέλω να θέσω μια ερώτηση για το θέμα του παθολογικού τζόγκου. Μπορείτε να μας πείτε ποιος εθίζεται στα τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή πρόκειται για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, πρόκειται για τους νέους ή ξέρουμε ε, ποια ομάδα ανθρώπων εθίζεται. Και κάτι ακόμη. Αν ρωτήσετε τους ε, ίδιους τους εθισμένους, ε, τι θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Θα ήθελαν, παραδείγματο χάρη, να έχουν περιορισμένη πρόσβαση για να αποτραπεί ο εθισμός ή ποια άλλα μέτρα θεωρούν ότι θα μπορούσαν να ληφθούν για να αποτραπεί ο εθισμός. Μάλιστα. Δηλαδή ρωτάτε σε τι συνίσταται ο παθολογικός τζόγος ή είπατε ποιος εθίζεται. Ε, κοιτάξτε, ο μέσος όρος των ανθρώπων που έρχονται ε, περισσότερο στα κέντρο μας έχουν ε, μέσο όρο ηλικία περίπου 25 για τους άνδρες, λίγο μεγαλύτερες είναι οι γυναίκες στην ηλικία. Αν δούμε τα δεδομένα, βλέπουμε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους άρχισαν να τζογάρουν πάρα πολύ νωρίς, κάποιοι και από 12 ετών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ε, όσο νωρίτερα ξεκινήσουν να παίζουν οι άνθρωποι τόσο πιο πιθανό είναι να εθιστούν αργότερα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Και Θέλω να προσθέσω ότι χρειαζόμαστε πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Εγώ με όλο ένα και περισσότερο που στην νομοθεσία στη Δανία ποτέ δεν έχει καλυφθεί το θέμα της πρόσβασης. Τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί εγώ στον τομέα αυτό μπορώ να σας πω ότι είναι πιο φθηνό να προλάβει κανείς παρά να θεραπεύσει και είναι και καλύτερο και από ηθική σκοπιά. Δηλαδή, τώρα λέτε τι χρειάζεται ε, για την πρόληψη, για να αποτραπεί ο εθισμός. Αν ρωτήσετε τους τι θα σας πούν. Πρόληψη χρειάζεται. Τα σχολεία μπορούν ε, να αφιερώσουν παραδείγματος χάρη μαθήματα για την πρόληψη του καπνίσματος ή μιλάμε για ασφαλή σεξουαλική ζωή αλλά δεν προσφέρεται κανένα μάθημα για τα τυχερά παιχνίδια. Το, κέντρο, το ερευνητικό κέντρο για την νεολαία στην, στην Δανία έκανε μία μελέτη για νεαρούς ανθρώπους γύρω στα 14 ως τα 16 έτη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραδείγματο χάρη και διαφήμιση επηρεάζει πάρα πολύ του νέου και ξέρουμε ότι το πόκερ, το οποίο είναι ένα σπορ ε, μάτσο, οδηγεί και στην ε, ανάπτυξη τέτοιου φαινομένου και χρειάζεται να έχουμε διαφήμιση και εκστρατεία κατά αυτών των φαινομένων. Να έχουμε λοιπόν πρόληψη και στα σχολεία και στον ε, υγειονομικό τομέα. Υπάρχει τεράστια ζήτηση Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ε, να έχουμε μία πρόληψη που θα διαρθρώνεται σε τρία-τέσσερα έτη. Αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει και τις ε, χώρες όπου υπάρχει κύριο αυτό το φαινόμενο, αλλά και όλη την Ευρώπη. Θα καλέσω και τους υπόλοιπους ομιλητές να απαντήσουν σε αυτό. Ο κύριο Μπρέκλα, αλλά και τον κύριο Ντέιβι θα καλέσω, αλλά και τον κύριο Μορέγη επίσης να απαντήσουν. Παρακαλώ, κύριο Σπεράκηλα, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να απαντήσω. Δεν ναι, νομίζω ότι κανείς θα ήταν κατά του γεγονότος ότι χρησιμοποιούμε τεχνικές δυνατότητες προκειμένου να περιορίσουμε τις ζημίες και αν ε, δεν ε, μπορούμε να προσδιορίσουμε παρκώς την ταυτότητα ενός ανθρώπου, τότε θα πρέπει να έχει κατώτερο πιστοτικό όριο, παραδείγματο χάρη, το άτομο αυτό. Και αν μπορέσουμε να το ταυτοποιήσουμε 100% τότε ε, θα μπορούσε να έχει πιο υψηλό πιστοτικό όριο. Θα πρέπει να υπάρχει, παραδείγματο χάρη, και ένα εθελοντικό εργαλείο να χρησιμοποιούν οι παίκτες, μπορούν να θέτουν ίσως και όρια στον εαυτό τους. Τώρα, ο επιγραμ, το επιγραμμικό, ο επιγραμμικός τζόγος, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια, ε, βλέπουμε ότι αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Υπάρχουν συναλλαγές όλο ένα και περισσότερες κάθε δευτερόλεπτο. Και ε, πολλές φορές δίνονται για κάποια εικονικά μπόνους παραδείγματος χάρη στους παίκτες και θα έπρεπε αυτά να απαγορευτούν. Ο κύριος Ντέιβιτ. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω ως εξής. Τώρα, η ίδια η φύση των τυχερών παιχνιδιών και του εθισμού στον τζόγο αποκαλείται συνήθως ε, κρυφός εθισμός και αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους αυτούς να συνεχίσουν να είναι εθισμό, εθισμένοι. Ανέφερε ο συνάδελφος ε, Γιώρσελ ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι ξεκινούν να παίζουν πάρα πολύ νέοι και μπορούν να το κρύψουν για πάρα πολύ καιρό. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ότι ε, κάποιο εμφανίζει τον εθισμό περίπου στα 45 του έτη, δηλαδή μπορεί να παίζει για 20-30 χρόνια χωρίς κανείς να το ξέρει. Και έτσι λοιπόν το να το αναφέρουμε αυτό ανοιχτά στην κοινωνία και να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία γενικώ για τους κινδύνους που ενέχουν τα τυχερά παιχνίδια είναι μια προσέγγιση. Πρέπει να δούμε τι επιτρέπει στον εθισμό να παραμείνει κρυφός και τι επιτρέπει στο άνθρωπο, στο άτομο, να συνεχίζει να τζογάρει. Και ένα από αυτά είναι η πρόσβαση. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα της πρόσβασης. Επίσης τα χρήματα επίσης και ο χρόνος. Γιατί ε, ακούτε να λέει κάποιος, α, Βαριέμαι. Δεν έχω καμία άλλη δραστηριότητα. Θα παίξω τυχαία παιχνίδια. Έτσι λοιπόν πρέπει να τα δούμε τα θέματα αυτά και σε κοινωνικό επίπεδο και να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα αυτό και ποια είναι τα συμπτώματα του εθισμού. Γιατί παραμένει κρυφός ο εθισμός. Δεν μπορεί, παραδείγματο χάρη, να κοιτάξει κάποιο έναν άνθρωπο και να πει «Α, έχει πρόβλημα, είναι εθισμένο στα τυχερά παιχνίδια. Ενώ στο διαδίκτυο, παραδείγματο χάρη, μπορεί κάποιο να δει πόσο χρόνο αφιερώνει ο παίκτη στα τυχερά παιχνίδια, τι ποσά ξοδεύει. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμπεριληφθούν στο σύστημα και παραδείγματο χάρη μπορούν να γίνει στέλνονται κάποιε υπενθυμίσει όταν χάνονται οι άνθρωποι αυτοί στον τζόγο. Δηλαδή πρέπει να δούμε γιατί παίζουν αλλά και τι γίνεται στο διαδίκτυο. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές ε, το διαδίκτυο και τα τυχερά παιχνίδια ως ε, διαφυγή. Έτσι λοιπόν ε, μπορούμε παραδείγματο χάρη να υπάρχει ένα ρολόι στην άκρη της οθόνης και κάποια στοιχεία να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί α, τόσο χρόνο έχω ξοδέψει παίζοντας, τόσα χρήματα και να έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα. Ναι, ο κύριο ε, Γιώργο Ελπρότεινο, ίσω εσεί και η Δανία μπορείτε να συνεργαστείτε. Κάθεστε και δίπλα-δίπλα, ξεκινήστε από σήμερα. Ναι, ε, κοιτάξτε, ένα μέλος της Γκαμπ έκανε ε, μια έρευνα για ε, το πώ παίζουν τυχερά παιχνιδιά οι νέοι και σίγουρα θέλουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίε και ίσω να εργαστούμε επί ενό project γιατί το έχουμε και εμεί αυτό το πρόγραμμα κατά νου, Κυρίω θέλουμε να εργαστούμε με του νέου. Ναι, επομένω, βεβαίω πρέπει να συνομιλήσουμε και οποιοδήποτε άλλο φυσικά θέλει να συνομιλήσουμε, ευχαρίστω. Ναι, νομίζω και οι δυο σα ε, θα ωφεληθείτε. Λοιπόν, κύριε Κενή, ξέρω πώ ήθελε να παρέμβει. Α ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μωρέη. Η κυρία Κιονή, την οποία πρέπει να έχω καλωσορίσει, είναι η συγκήτρια για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων. Κύριος Μωρέη, πρώτα απ' όλα. Ναι, σύντομα. Προφανώς δεν είμαι ο ειδικό ε, στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω όμως πως ε, οι αθλητικές οργανώσεις έχουν ένα ρόλο να παίξουν όσον αφορά τη χορηγία, τις διαφημίσεις. Ε, εμείς αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε ένα κώδικα συμπεριφοράς για τους συλλόγου μας ε, που αφορά εμπορικές ε, συμφωνίες ε, με εταιρείε στοιχημάτων για να τηρούνται κάποιες βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφήμιση και την ασφάλεια των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο. Ας ακούσουμε την κυρία Οκινή που ήθελε να κάνει κάποια σχόλια ή ερωτήσεις να σας ακούσουμε για λίγο χρόνο. Ευχαριστώ και θα είμαι σύντομη. Ε, ζητώ συγγνώμη, έφτασα αργοπορημένη, αλλά είχαν λυμμένες υποχρεώσεις. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Άκουσα παρόλα αυτά ένα κομμάτι τη συζήτηση και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ε, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι όλοι οι ομιλητέ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που άκουσα. Θα ήθελα να θέσω ένα επιπρόσθετο ερώτημα γιατί υπόθηκαν τα περισσότερα ήδη ή μάλλον μια διευκρίνηση θα ζητήσω από τον κύριο Μοχέγε μίλησε για την ε, γεννήκευση των συμβατικών σχέσεων ανάμεσα στους φορείς εκμετάλλευσης και τους διοργανωτές των αθλητικών εκδηλώσεων. Τι εννοεί ε, μιλώντας για αυτές τις ε, συμβατικές σχέσεις, μιλάτε για την αναδιανομή ε, κερδών και αν ναι, υπό ποια μορφή. Μάλιστα, ευχαριστώ για την ερώτηση. Προσπάθησα να το εξηγήσω και εγώ και ο κύριος Βιλότε εξάλλου. Αυτό το θέμα των συμβάσεων και των νομικά δεσμευτικών ε, σχέσεων ε, έχει κέρια σημασία για να υπερασπιστούμε την ακυριότητα του ήθος στο χώρο του αθλητισμού. Τι εννοώ λοιπόν. Οι αθλητικές ενώσεις θα πρέπει, ε, μάλλον θα πρέπει να ακουστεί η φωνή των αθλητικών ενώσεων υπό την αιγίδα, υπό τον έλεγχο αν των εθνικών αρχών σε σχέση με την προσφορά στοιχημάτων για τις δικές τους εκδηλώσεις. Θα προσπαθήσω να διευκρινίσω αυτό που εννοώ. Absolument αυτοί που κατέχουν τα δικαιώματα για την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων ε, δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ε, οργανώσεις ε, στοιχημάτων προσφέρουν στοιχήματα για τις δικές μας αθλητικές εκδηλώσεις χωρίς καν να μας ενημερώσουν, χωρίς να ενημερώνουν για τη ροή χρημάτων, για τα ποσά που έχουν στοιχηματιστεί, για το είδος των στοιχημάτων, για τους κινδύνους που συνδέονται λόγω κάποιων κωδίκων ε, υπάρχουν προγράμματα που έχουν εφαρμόσει ήδη οι φορείς εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς. Θεωρούμε ότι είναι θετικές οι κινήσεις. Τούτου λεχθέντος ε, εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα ε, της μη επικοινωνίας, μη συστηματικής επικοινωνίας με τους φορείς εκμετάλλευσης. Για να έχουμε μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στους διοργανωτές των αθλητικών εκδηλώσεων και το, τους φορείς εκμετάλλευσης που ουσιαστικά οργανώνουν μια εμπορική δραστηριότητα που φέρει επί των αθλητικών συναντήσεων χωρίς να μας ενημερώνουν, χωρίς να ενσωματώνουν στην απόφαση για αυτή τη συμβατική σχέση. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχουν αναλυφθεί κάποια μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το μοντέλο υπάρχει και στην Αυστραλία και σε κάποιες άλλες χώρες. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα σε περισσότερες χώρες, ε, ε, μιλώντας για την αναδιανομή κερδών. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα τζακ πότε. Είδατε τα στατιστικά στοιχεία για τη Γαλλία. Πόρο απέχουμε από αυτό. Είναι, τίθεται πραγματικά ζήτημα ηθικής. Ε, και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας ακούσει και να προτείνει να υπάρξουν απλώς συμφωνίες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τελειώσει και αυτή η τελευταία συνεδρία μας και να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα και βεβαίως καλό θα είναι να παραμένετε σε επαφή μαζί μας και νομίζω πως και η Κομισιόν θα θέλει να ε, έρθει σε επαφή μαζί της. Οπότε θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την κυρία Μπρόμπτε να κάνει κάποια σχόλια. Είναι αρμόδια τώρα για το θέμα αυτό στη Γενική Διεύθυνση Ιστορικής Αγοράς και ε, θα ήθελα να της δώσω το, το λόγο να μας πει κάποιες σκέψεις ε, για αυτά τα οποία ακούστηκαν και μετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κρόιτσμαν. Σας ακούσουμε πρώτα την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω όσα είπατε μόλις ότι αυτή η ακρόαση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και για την Κομισιόν. Πρόκειται για στοιχεία που θα λάβουμε υπόψη στην ευρύτερη διαβούλευση που ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε μια σειρά σημείων όπου συγκλίνουν οι συμμετέχοντες διαπιστώνουμε καταρχήν ότι τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλο βαθμό ευκαιρία στην οργάνωση των εθνικών του συστημάτων, αλλά όποιο και να είναι η φύση των συστημάτων αυτών, όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν το ίδιο φαινόμενο με διαφορετική ένταση φυσικά, παράνομα φαινόμενα που προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει νομίζω ένα διακύβευμα σε κοινοτικό επίπεδο για να εξετάσουμε ποιο είδους παρέμβαση και πρόσφατης βοήθειας ε, θα χρειαστεί έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά αυτά τα παράνομα φαινόμενα. Και το ερώτημα είναι ακριβώς το εξής, πώς μπορούμε να το πράξουμε. Είχαμε και συζητήσει και στο Συμβούλιο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τα κράτη-μέλη επίση συζήτησαν το θέμα αυτό. Και είναι αλήθεια ότι η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των αριθμιστικών αρχών είναι ένα θέμα το οποίο σε επίπεδο Συμβουλίου φαίνεται ότι την χάνει ευρεία ε, συμφωνία Τώρα το θέμα είναι να ξέρουμε τι θα εννοούμε με την έννοια διοικητική συνεργασία και μέχρι πού μπορούμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πιθανότατα ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξή, ότι η συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και κρατών μελών δεν μπορεί να γίνει χωρί να υπάρχει μία ελάχιστη συμφωνία για τα είδη των πληροφοριών που θέλουμε να ανταλλάξουμε και επίση ε, για τους λόγους για τους οποίους θέλουμε αυτή την ανταλλαγή των δεδομένων. Δηλαδή να υπάρχουν κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και να εξετάσουμε σε σχέση με τους λόγους με τους οποίους υπάρχει παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών. Αναφέρθηκαν ε, εδώ σήμερα το θέμα του ήθους, ε, η προστασία των παικτών, πολέμηση, της νομοποίησης των παράδομων εσόδων. Υπάρχουν ε, δηλαδή πολλοί λόγοι για την προστασία των καταναλωτών αλλά και τη διατήρηση της δημοσίας τάξης για να πέμβουν οι ρυθμιστικές αρχές. Εμείς λοιπόν θεωρούμε προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε φυσικά είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση και σήμερα είδαμε και από τον αριθμό των συμμετεχόντων θα έχουμε πολλές απαντήσεις φανταζόμαστε στην πράσινη βίβλο και τον Αύγουστο θα αρχίσουμε να αναλύουμε αυτές τις απαντήσεις έτσι ώστε το φθινόπωρο να μπορέσουμε να εκπονήσουμε μία έκθεση κατόπιν της διαβούλευσης και φυσικά κατανοούμε ότι και το Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει την έκθεσή του πριν ολοκληρώσει η Κομισιόν τις εργασίες της στο θέμα αυτό έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη το σύνολο των δεδομένων και των συζητήσεων που θα έχουν λάβει χώρα και στη δική σας επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και βεβαίως αναμένουμε τη συνεργασία μας στο σημαντικό και ενδιαφέροντα θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για να ολοκληρώσει και τον ευχαριστώ που οργάνωσε αυτή την ε, ακρόαση και βεβαίως φρόντισε να βρει τόσο πολλούς και διακεκριμένους ομιλητές. Κύριε Κρότσιμα, αν έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ και τους και οδησηγητές που έκαναν τις προτάσεις τους σε μια συνάντηση και ε, προσπαθήσαμε να καλύψουμε το θέμα πανευρωπαϊκά και να περιοριστούμε σε μια χώρα. Συνοψίζοντας, οι απαιτήσει που ακούστηκαν ήταν καταπολέμηση του παρανόμου παιχνιδιού, καταπολέμηση της απάτης, καταπολέμηση της εξάρτησης. Είδαμε τι κάνει η Φιλανδία με την άδεια πρόσβασης. Που ε, πλέον ε, βλέπουμε πως τα πράγματα ζητάνε ευρωπαϊκή ρύθμιση. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε και την αρχή της επικουρικότητας. Και τώρα θα είναι συναρπαστικό να δούμε το τι θα έχουμε. Γιατί με τους ε, σκιώδει ε, εισηγητέ. γιατί βεβαίω η πράσινη βίβλο τα αφήνει όλα ανοιχτά. Οπότε αν υπάρχει ευρεία πλειοψηφία στο κοινοβούλιο μπορούμε να ασκήσουμε κάποια πίεση στα κράτη-μέλη βεβαίω να συνεργαστούν περισσότερο γιατί νομίζω πως όλες οι ομάδες θέλουν κάτι τέτοιο, οι κοινοβουλευτικές ομάδες και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την αρχή της επικουρικότητας. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να κάνουν κάτι, αλλά εάν δεν κάνουν και τίποτα θα έχουμε κατακαιρματισμό που δεν θα προσφέρει τίποτα. Και νομίζω πως πραγματικά μόνο μέσω ευρωπαϊκής ρύθμισης μπορούμε να λύσουμε αυτό το, το πρόβλημα. σεβόμενοι όπως είπα την αρχή της επικουρικότητα. Δεν ξέρω, θα μπορέσουμε να βρούμε μια διατύπωση, να ζητήσουμε κάτι από την Κομισιόν να προχωρήσει το, το θέμα. Νομίζω και η κυρία Σαλτεμόζε συγκατα... συγκατένευσε. Νομίζω λοιπόν πως ε, δεν θέλουμε να ε, καταλήξουμε χωρίς αποτέλεσμα. Οπότε θα προσπαθήσουμε εγώ και οι σκιώδεις συζητητές να επιτύχουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνοντας, να σας πω το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Κρότσμα θα στείλει την έκθεση για μετάφραση την ερχόμενη εβδομάδα. 12 Ιουλίου θα την εξετάσουμε στην Επιτροπή, 18 Ιουλίου προθεσμία για τροπολογίες, θα τις δούμε τον Αύγουστο, μετά τις τροπολογίες θα ψηφίσουμε τον Σεπτέμβρη. Και νομίζω αυτό ταιριάζει και με το πρόγραμμα της Κομισιόν για την εξέταση των απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο. Οπότε ευχαριστώ τους συμμετέχοντες ακόμη μια φορά. Νομίζω αξίζουν ένα χειροκρότημα. Uh, thank you very much. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω στα μέλη της Επιτροπής ε, πως ε, ξαναρχόμαστε εδώ πέρα αύριο το πρωί στις 9 με τον Ούγκρο Υπουργό Ανταγωνιστικότητας, τον κύριο Σέφελ που με καλός φίλος της Επιτροπής θα μας πει τα της Ουγγρικής Προεδρίας. δέκα η ώρα μετά θα εξετάσουμε την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και μετά μια άλλη ενδιαφέρουσα ακρόαση για το μέλλον της ελληνικής πολιτικής με τον κύριο Σαλβίνη και νομίζω πως η κυρία Σαλντεμόζε θα ξαναέρθει, ελπίζω να ξαναέρθει γιατί και με αυτό το θέμα ασχολείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σας βράδυ.